Okay. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, on aimerait commencer. Καλησπέρα σας. Να αρχίσουμε. Ich werde auf Deutsch sprechen. Θα μιλήσω γερμανικά. Yeah. Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί συμμετέχοντες, χαίρομαι όλο ιδιαίτερος που σας καλωσορίζω στην τρίτη μας συνεδρία για σήμερα που αφορά τη διευκόλυνση της ζωής των πολιτών της Ευρωπαϊκής συγκεκριμένα στο στα δικαι... σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και των γονέων ε, διότι όλο και περισσότεροι κινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την μετακίνηση αυτή προς ένα άλλο κράτος μέλος ε, συνδέεται και ε, η οικογενειακή σχέση και έχοντας περισσότερους διασυνοριακούς γάμους έχουμε και περισσότερα διασυνοριακούς συνοριακά διαζύγια και χωρισμούς οικογενειών. Όταν λοιπόν έρχεται ένα μέλος της οικογενείας και ακολουθεί το ένα γονέα ενδέχεται να ζουν σε διαφορετικά ε, κράτη γονείς και δημιουργούνται προβλήματα ιδίως με το δικαίωμα επίσκεψης οπότε μπορεί να οδηγήσει αυτό στην απαγωγή ενός παιδιού από τον ένα γονέα και αυτό είναι ένα συνεχές ε, πρόβλημα διότι και οι γονείς και τα παιδιά υποφέρουν ε, εξίσου και έχουμε ήδη προχωρήσει σχετικά ε, με την με ε, ε, το θέμα των ε, επισκέψεων των παιδιών υπάρχει μια χάρτα των δικαιωμάτων του παιδιού και λέγεται ότι το παιδί έχει δικαίωμα για τακτικές σχέσεις και με τους δύο γονιούς για να μπορέσει να ευημερήσει και υπάρχει ένας κανονισμός σχετικά με την λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή των δικαστικών δικαστικών ε, αποφάσεων σχετικά με ε, την γονική κατάσταση. Υπάρχει μία αυτόματη αναγνώριση του δικαιώματος επίσκεψης σε όλα τα κράτη αλλά στον κανονισμό αναφέρεται επίσης ε, και η δυνατότητα τα παιδιά να μπορούν να αναπτυχθούν ομαλά και συγχρόνως αποφεύγουμε έτσι τις απαγωγές παιδιών και από το έχουν ρυθμιστεί τα αστικά θέματα της προστασίας του παιδιού και αποφυγή των απαγωγών και το θέμα αυτό έχει πραγματευτεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε έναν διαμεσολαβητή για τις διασυνοριακές απαγωγές των παιδιών. Έχουμε ε, την κυρία Αντζελίλη, αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι υπεύθυνοι για το θέμα αυτό για να μπορεί να υπάρχει μια ελεύθερη επικοινωνία και μεταξύ των δύο γονέων κατά τρόπον ώστε να ε, είναι το καθεστώς αυτό προς όφελος του παιδιού και έχουν διατυπωθεί πολλές προτάσεις για αποφυγή των απαγωγών παιδιών και αυτό η απάντηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει κάνει διάφορα ψηφίσματα και στη συνέχεια μία μελέτη για τα δικαιώματα των γονέων και την ε, ε, ρύθμιση των ε, επισκέψεων των γονέων κατά τρόπον ώστε να μπορέσει να ρυθμίσει θέματα που δεν κατάφεραν να ρυθμιστούν στα εθνικά δικαστήρια από τον δυσαρεστημένο γονιό. Τονίζονται ορισμένα θέματα και σήμερα θα μας παρουσιαστούν ορισμένα αποτελέσματα των προσπαθειών μας. Έχουν γίνει μεγάλες ε, ε, μεγάλες ε, πρόοδοι αλλά πρέπει να ρυθμίσουμε αυτό το θέμα και να το προσαρμόσουμε στα νέα, στα νέα καθεστώτα που διέπουν τις οικογένειες. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να συμπληρώσει τα δικαιώματα μητρότητος ε, για να ε, μπορεί ε, να, ένας γονιός να αναγνωρίσει το δικαίωμά του σε ένα άλλο κράτος μέρος, να γράψει το παιδί στο σχολείο και δεν είναι αυτόματη αυτή η αναγνώριση στα άλλα κράτη-μέλη. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι και οι δύο πλευρές και οι γονείς και τα παιδιά πρέπει να έχουν νομική ασφάλεια και ε, ε, το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων έχει αναφερθεί και εις τις διασυνοριακές υιοθεσίε που θα θυγούν σήμερα. Θα ήθελα να πω κάτι ακόμη ε, σχετικά με την μητρότητα και την, τις βιολογικές μητέρες διότι υπάρχουν πλέον μέθοδοι για να ικανοποιηθούν οι οικογένειες που δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά αλλά αυτό οδήγησε σε νομικά προβλήματα δηλαδή την αναγνώριση του δικαιώματος του γονέα και την υπηκότητα του παιδιού. Πρέπει λοιπόν να ρυθμίσουμε και αυτά τα θέματα και να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στις ευρωπαϊκές οικογένειες να ζουν αξιοπρεπώς. Θέλω να ευχαριστήσω ε, την ε, διπλανή μου ε, η οποία θα παρουσιάσει τις μελέτες της και συγχρόνως θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ρομπέρτα Αντζελίλη η οποία είναι αντιπρόεδρος του Ιδρύματος κατά των απαγωγών των παιδιών και τους ομιλητές στους οποίους θα δώσω το λόγο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να περιοριστείτε στο χρόνο των 10 λεπτών για να έχουμε στη συνέχεια επαρχή ε, χρόνο για να συζητήσουμε και μου έχουν δοθεί οδηγίες να σέβομαι ακριβέστατα το χρόνο. Τώρα λοιπόν θα, θα κάνουμε ε, την ε, συζήτηση του πρώτου θέματος, δηλαδή την κατάσταση με την εφαρμογή των Βρυξελών 2, του κανονισμού Βρυξελών 2, ιδίω όσον αφορά την διασυνοριακή εφαρμογή ε, των αποφάσεων σχετικά με τα παιδιά. Η παρουσίαση θα γίνει από τον Τζαν Παόλο Ρωμάνο, που ε, θα παρουσιάσει τη μελέτη ενός Ελβετικού Ινστιτούτου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ο φορέας που εκπροσωπώ κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει μια μελέτη για τη γονεϊκή ευθύνη απέναντι στα παιδιά, για την γονεϊκή επιμέλεια και τα δικαιώματα επίσκεψης πέραν των συνόρων. Η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο, βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ ε, το τμήμα που διοργανώνει αυτή την ημερίδα προβληματισμού. Είναι ο προνομιούχος μας συνομιλητής στην διάρκεια αυτού του προβληματισμού που στόχο έχει να κάνει τον απολογισμό των προβλημάτων, των πρόοδων που έχουν σημειωθεί και των πιθανών μελλοντικών λύσεων. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιους από τους καρπούς αυτής της έρευνας. Καταρχήν, δεν αμφιβάλλει κανείς ότι ο κανονισμός ε, Βρυξέλλες 2α έφερε ένα σημαντική πρόοδο ε, πάνω στο θέμα που αποτελεί και τον τίτλο αυτής της ημερίδας, την απλοποίηση της ζωής των πολιτών. Θα σας περιγράψω σε γενικές γραμμές τα προβλήματα. Η αρχή είναι ότι συνήθως είναι υπεύθυνο και αρμόδιος ο δικαστής της συνήθους διαμονής του παιδιού, απόφαση 10 Απριλίου του 2010. Ε, αυτό μεταφράζει ε, την ένταξη του παιδιού σε ένα ορισμένο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον και έχει συγκεκριμενοποιηθεί αυτή η προστασία μέσα από μια σειρά δικαστικών αποφάσεων. Επομένως ε, ε, μπορούν να, υπάρξουν και κάποιες παρεκκλήσεις και να υπάρξει κάποια δικαστική μεταφορά και ανταλλαγή αρμοδιοτήτων και δοσιδικίας. Η γερμανική και η γαλλική νομολογία δείχνει ότι αυτή η ανταλλαγή πολύ συχνά ζητείται από το ένα μέλο από το ένα μέρος, από το ένα ένδικο μέρος. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Και πάλι η εθνική νομολογία δείχνει τη χρησιμότητα αυτής της παρέκκλησης γιατί πάντοτε αποβαίνει υπέρ του ε, δικαστή του διαζυγίου ή του εθνικού δικαστή του παιδιού μια απόφαση που μπορεί μια απόφαση, ε, αυτό κρίθηκε με μια απόφαση εφετείου της Πολωνίας Όσο αφορά την αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων, αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών διαδικασιών. Ε, υπάρχει μια σειρά αιτιολογήσεων απόρριψης της εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης και ε, έχει απλοποιηθεί η διαδικασία εκτέλεσης των ε, αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων σε παραπέμπω στον αριθμό 44. Ο κανονισμός αυτός προβλέπεται από την συνθήκη της Χάγης και το πιο το πιο... η πιο ενδιαφέρουσα όψη είναι η σύγκρουση μεταξύ των αποφάσεων μη επιστροφής και της απόφασης που επιβάλλει την επιστροφή με βάση το... την χώρα διαμονής. Η απόφαση επιστροφής πρέπει να πιστοποιηθεί φυσικά και ο εκτελεστός τίτλος εκδίδεται στον ευρωπαϊκό χώρο. Η σημασία αυτής της διάταξης έχει υποστηριχτεί θερμά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις μεγάλες σχετικές υποθέσεις. Πέρα από αυτό, οι αποφάσεις που αφορούν τα δικαιώματα επίσκεψης ε, επίσης πιστοποιείται και επενδύεται την, ε, την ισχύ εκτελεστού τίτλου. Ποιος είναι ο απολογισμός λοιπόν τώρα με βάση τον εθνικό, την εθνική νομολογία. Μετά από έξι χρόνια εφαρμογής του κανονισμού Βρυξέλλες 2α, μάλλον θετικός είναι ο απολογισμός υπήρξαν κάποιες δυσκολίες εφαρμογής που επιλύθηκαν πολλές φορές από την εσωτερική νομολογία γιατί το ευρωπαϊκό δικαστήριο δεν θα μπορούσε να τις επιλύσει. οκτώ αποφάσεις έχουν δει το φως και ανοίγουν μια πολλά υποσχόμενη οδά. υπάρχει ένα σύστημα προστασίας των γονεϊκών δικαιωμάτων ε, ε, βελτιώνεται η προστασία τους και θα σας παρουσιάσω ε, τέσσερις πτυχές. πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά τη γονική επιμέλεια, οι λόγοι απόρριψη τη αναγνώριση είναι πολύ άριθμοι. Το άρθρο 23 του κανονισμού απαριθμεί 7 τέτοιου λόγου. Και αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στην ε, δικαστική ανθολογία για να δούμε ε, ότι πολύ σπάνια είναι συμπαθητική η απόρριψη αυτής της αρμοδιότητας. Από το Σλέχης Χόλσταϊν το δικαστήριο αρνήθηκε να αναγνωρίσει ε, μια απόφαση του δικαστηρίου ανηλίκων του Μιλάνου που είχε να κάνει με την γονική επιμέλεια ως λόγος άρνησης. Ε, έτσι με αυτόν τον λόγο άρνησης ανοίγει μια σειρά αποφάσεων που χρειάστηκε να επανέλθουν και να εκδώσουν καινούρια δικαστική απόφαση διαφορετική από αυτή που είχε εκδοθεί στην αρχή. περίπτωση ε, σύγκρουσης μεταξύ δικαστικών αποφάσεων ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες όπως ξέρετε. Πριν από λίγες εβδομάδες ε, βγήκε και μια καινούργια απόφαση εφετείου που το αποδεικνύει. Έχουμε την οικοδόμηση λοιπόν ενός χώρου ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης, ο οποίος υποστηρίζεται έτσι η γερμανική απόφαση δίνει το παιδί στη Γαλλία, η απόφαση του Γαλλικού Δικαστηρίου δίνει το παιδί στη Γερμανία και το παιδί βρίσκεται χαμένο. Ε, ο γονέας που έχει εξουσίες πάνω στο παιδί λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για τα θέματα υγεία, σχολείου κτλ. Αυτό οδηγεί σε μια πραγματικά άρνηση απονομή δικαιοσύνη σε κοινοτικό επίπεδο. Πράγμα που προφανώ είναι αντίθετο με τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελεί και εμπόδιο στην πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Από ό,τι φαίνεται ο κανονισμός έχει δύο πρόσθετους μηχανισμούς για να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Υπόθηκε και το πρωί από την κυρία Επίτροπο Ρέντινγκ την επέκταση ενός μηχανισμού αναγνώρισης σε όλες τις αποφάσεις για την γονική ευθύνη και μέρημνα μιλάμε για δικαιώματα πιστοποιημένα για τα δικαιώματα επίσκεψης των γονέων. Τα ανέπτυξαν οι συνάδελφοι. Νομίζω ότι αυτός ο διπλός μηχανισμός διαφέρει, αυτός ο διπλός μηχανισμός θέλει να Υπάρχει μια πτυχή για τα δικαιώματα επίσκεψης, μια πτυχή για τα δικαιώματα γονικής μέρημνας ε, και, προσπαθούν οι δύο αυτοί μηχανισμοί να εγκαταστήσουν έναν ενοποιημένο ομαλό μηχανισμό, ενιαίο μηχανισμό αντιμετώπισης των θεμάτων. Έχουμε ένα σύστημα που μας λείπει. Δεν έχουμε σύστημα επίλυσης σύγκρουσης αποφάσεων. Ε, μπορούμε να σκεφτούμε τι είδους συγκρούσεις προκύπτουν και ίσως θα έπρεπε να συσταθεί μια ειδική σύνθεση δικαστηρίου για να δικάζει τις, τις οικογενειακές αυτές υποθέσεις. Έπειτα, δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ δικαστών για την χορήγηση, της, την της, την επιδίκαση της γονικής μέρημνας στις διασυνοριακές διαφορές οι δύο γονείς μπορεί να μένουν σε διαφορετικές χώρες και μπορεί να έχουν σημαντικές επαφές με το παιδί, αλλά ποιος έχει αρμοδιότητα να κρίνει σε περίπτωση διαφοράς. Ε, ένας είναι ο δικαστής που θα κρίνει. Ο εθνικός δικαστής δεν είναι κατά ανάγκη ο πιο εξοπλισμένος για να καλύψει αυτήν την περίπτωση γιατί η οπτική θέση παρατήρησης είναι μεροληπτική. Είναι δύσκολο να αποφύγουμε να έχουμε μια Ιταλογερμανική κατάσταση για να πάρουμε ε, την ε, υπόθεση που, για την οποία χύθηκε περισσότερο μελάνι τι γίνεται όταν το παιδί προσυδειάζει πιο πολύ στα συμφέροντα του γερμανικού κράτους. Τι, τι γίνεται εκεί πέρα. Νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή μπορούμε να δώσουμε στο δικαστή τη συνήθους διαμονής του άλλου γονέα τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις αν μη τι άλλο, δηλαδή να κάνει μια εκτίμηση για το συμφέρον του παιδιού. Ή από την πλευρά της Ιταλίας, ο δικαστής της συνήθους διαμονής, ο Γερμανός για παράδειγμα, θα μπορούσε να λάβει υπόψη στην αιτιολογία του τις τυπικές αποφάσεις του, της γερμανικής μεν πλευράς, αλλά με την ιταλογερμανική τους διάσταση έτσι ώστε να μπορεί και ο Ιταλός δικαστής να προσκομίσει και αυτό στοιχεία. Και έτσι να εκμεταλλευτούμε να, να εκμεταλλευτεί κανείς το δικαστικό δίκτυο που υπάρχει. Ο κανονισμός κατ' ουσίαν προβλέπει ήδη την δυνατότητα ενός τέτοιου δικαστικού διαλόγου. Υπάρχει ο, ο μηχανισμός του άρθρου 15 ε, που προκρίνει την ε, καλύτερη ε, δικαιοδοσία. Φτάνω στο τέλος του χρόνου που μου αναλογεί. Πολλής λόγος έγινε για το ε, δίκαιο, το εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο όσο αφορά και την ε, επιδίκαση της γονικής επιμέλειας. Υπάρχει και ο χωρισμός μη εγγαμών γονέων. Σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, η μητέρα αποκτά την αποκλειστική γονική επιμέλεια σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει μια συνθήκη, συνθήκη του 1996 της Χάγης. Η λύση αυτής της συνθήκης δεν μας φαίνεται σύμφωνη με τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί εκεί αφορά μόνο ε, τη δυνατότητα του γονέα να ορίζει εκείνος το εφαρμοστέο δίκαιο. Αυτό ίσως μπορεί να ισχύσει σε περιπτώσεις πολύ ξεκάθαρων συμφωνιών μεταξύ των γονέων. Αλλά πάντως το συμφέρον του παιδιού πρέπει πάντοτε να εξασφαλίζεται. Οι γονείς από τη γέννηση του παιδιού μπορούν να επιλέξουν για παράδειγμα την εφαρμογή του γαλλικού δικαίου που είναι πιο γενναιόδωρο σε περίπτωση χωρισμού υπάρχουν και τα συμπεράσματα της μελέτης τα οποία μπορείτε να δείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης. Αντιλαμβάνομαι ότι ε, υπάρχει ένας θετικός απολογισμός παρόλο που ε, δεν μπόρεσε το Διεθνές Δικαστήριο να ε, ρυθμίσει όλα τα θέματα θετικά. Και προτού φτάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως θα ήθελα να χαιρετήσω απαιτήσω εις ε, το θεωρείο των επισκεπτών μία ομάδα επισκεπτών του συναδέλφου Μάντερς και έρχομαι στο επόμενο θέμα που είναι το διασυνοριακό ε, διασυνοριακή άσκηση του δικαιωμάτου επίσκεψης από την κυρία Τόμα Τατβόκ από τη Βιέννη. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω μπροστά σε ένα πολυπληθές γερμανόφωνο κοινό. Θα ήθελα τώρα εδώ να εστιαστώ στην εφαρμογή του δικαιώματος επικοινωνίας. Δηλαδή τι κάνουν ε, τα δικαστήρια σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας και πώς μπορεί αυτό να χορηγηθεί ε, επιτυχώς. Είναι ένας πολύ ευαίσθητος χώρος αλλά είναι ένα βασικό δικαίωμα ε, της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών Λοιπόν, Ισχύει δύσκολα ήδη στο τομέα του εθνικού δικαίου. Όταν πρόκειται για διασυνοριακές σχέσεις τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Ο βασικός στόχος σε ε, πολυμερείς συμφωνίες είναι να ε, υπάρξει μία αποτελεσματική εφαρμογή στα μεμονωμένα κράτη. Στο οικογενειακό δίκαιο πρέπει κανείς να καταφεύγει όλο και περισσότερο ε, σε ε, ε, κοινοτική νομοθεσία για να ρυθμίσει τα πολιεθνικά προβλήματα και θα πρέπει να υπάρχει όλο και περισσότερο αναργόνηση των αποφάσεων, δημιουργία μηχανισμών και θεσμικών οργάνων που θα μπορέσουν να μεσολαβήσουν και να οργανώσουν τις διατυπώσεις για να εξασκηθούν το δικαίωμα της επίσκεψης. Ε, πού οφείλεται το πρόβλημα. Ε, οφείλεται διότι πρέπει να διατηρηθεί η επικοινωνία ε, παρόλο που ένας γονιός έχει μετακομίσει σε κάποια άλλη χώρα και πρέπει να σας πω τι δυνατότητες έχουμε για να επικαλεστούμε το θέμα, το δικαίωμα αυτό. Οι Βρυξέλλες η ε, γονική μέρημνα η οποία εδώ αναφέρεται ε, άπτεται και του δικαιώματος επίσκεψης και αναγνωρίζει ορισμένα εχέγγυα για, να, ε, για την εξάσκηση αυτού του δικαιώματος επικοινωνίας και επιπλέον έχουμε το ευρωπαϊκό δίκαιο και την απόφαση του δικαστηρίου για τα παιδιά όταν πρόκειται για το δικαίωμα επίσκεψης και επικοινωνίας. Το δεύτερο θέμα το οποίο θα ήθελα να επικαλεστώ είναι ότι διαπιστώνουμε ότι πρέπει συγχρόνως να διευκρινιστεί η διεθνής αρμοδιότης, δηλαδή ποιο δικαστήριο είναι υπεύθυνο. Είναι κάτι το οποίο έχει σχέση ε, με την εξάσκηση ενός δικαιώματος. Ο κανονισμός Βρυξέλλες 2 ε, επέλεξε ε, να θεωρήσει ε, σαν, ε, σαν τόπο συνήθους διαβιώσεως του παιδιού και σε περίπτωση όπου το παιδί αυτό μεταφέρεται σε κάποιο άλλο ευρωπαϊκό κράτος προβλέπονται ορισμένες διατυπώσεις για τους επόμενους τρεις μήνες. Γιατί, Γιατί έτσι μία δικαστική απόφαση του δικαστηρίου που έχει ασχοληθεί με το θέμα ε, καταρχήν πρέπει να μπορέσει να διατηρηθεί και ε, να υπάρξει μία προσαρμογή στην ε, τροποποιημένη κατάσταση. Ξέρετε ότι αν υπάρξει παράνομη κατακράτηση ενός παιδιού ή απαγωγή τότε συνεχίζουν να διέπεται από το ειδικό αυτό καθεστώς το παιδί επί έναν επιπλέον χρόνο και ε, ε, πρέπει να υπάρχει μια δικαστική απόφαση η οποία να εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες και δημιουργήθηκε στον κανονισμό Βρυξέλλες 2 ένας ευρωπαϊκός τίτλος επίσκεψη ο οποίος αποτελεί μία μεγάλη ε, εγγύηση. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην επικοινωνία του παιδιού πρέπει να καταρτίζονται βάσει του άρθρου 41 και να είναι άμεσα εκτελεστές χωρίς, χωρίς περαιτέρω αποφάσεις εκτελέσεως ή χωρίς να μπορεί να ανακληθεί η εκτέρεσή τους και συμφωνώ με ε, τον προλαλήσαντα ότι τα δικαστήρια δεν είναι πάντοτε πολύ σοφά σε αυτό το τομέα. Η, ε, εκτέλεση, η εκτέλεση της απόφασης είναι ένα βασικό θέμα και πρέπει να υπάρξει και ένας ε, έλεγχος ο οποίος ενδέχεται να ε, αποσιάζει τελείως. Πρέπει να υπάρχει μία διαδικασία η οποία υπό υπόκειται στον χώρο όπου διαμένει το παιδί και ε, εκεί μπορεί κανείς να ε, επικαλεστεί ε, την ε, παράνομη άρνηση επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα άλλο θέμα το οποίο όμως ρυθμίζεται διαφορετικά στα διάφορα κράτη-μέλη. Σε ορισμένα κράτη όπως η Αυστρία δεν υπάρχει υποχρεωτική αφαίρεση του σε περίπτωση που ο γονιός αρνηθεί το δικαίωμα επίσκεψης. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο δικαίω, δίκαιο επικοινωνίας και εις την ε, ε, απαγωγή του παιδιού διότι ε, το δικαίωμα επισκέψεως αφαιρείται μετά από μία απαγωγή ή ε, μετά την επιστροφή του παιδιού πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα της ε, επικοινωνίας με τον γονιό ο οποίος το είχε απαγάγει ή την ε, διακοπή της επικοινωνίας με τον γονιό από τον οποίο αφαιρέθηκε το παιδί. Σε όλα αυτά τα σημεία προκύπτουν πολλά προβλήματα αφενός όσον αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας στο Το δικαίωμα επικοινωνίας πρέπει να προσαρμοστεί σε μία ε, διαφορετική κατάσταση από πλευράς τόπου αλλά να μην υπάρξει μία διακοπή της ε, επαφής η οποία μπορεί να υπάρξει εάν ληφθούν ε, στα γρήγορα αποφάσεις. Παραδείγματος χάρη ποιο είναι το κόστος ταξιδίου. Ενδέχεται να χρειαστεί οικονομική βοήθεια οικογένεια και δέχεται να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικέ μέθοδοι παραδείγματο χάρη διεθνή διαμεσολάβηση για να μπορέσουν να υπάρξουν επαφές για να αποφευθεί η διακοπή της επαφής και ε, για να αποτραπούν οι παρανοήσεις και ε, οι διαφορές. Επίσης, σε σχέση με μία παγωγή ενός παιδιού διαπιστώνουμε ότι υπάρχει φόβος του παιδιού, του γονιού ότι θα υπάρξει και περαιτέρω απαγωγή και κατόπιν αυτού άρνηση επικοινωνίας οπότε δεν θα μπορούν ενδεχομένως να υπάρξουν ε, επισκέψεις με κάποια συνοδεία. Ως εκ τούτου η αρμεδιότης του δικαστηρίου παραμένει η στο αρχικό κράτος για το δικαίωμα επικοινωνίας και επαφής. Αλλά συγχρόνως υπάρχει και αρμοδιότητα του δικαστηρίου του νέου κράτους όπου διαμένει το παιδί και πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη. Στο θέμα της ε, αποφάσεως για το δικαίωμα επικοινωνίας πρέπει να συνυπολογιστούν όλα αυτά τα θέματα. Έχουμε ε, μία περίπτωση ε, όπου ο ένας γονιός ήταν Γερμανός και ο άλλος Ιταλός και που απασχόλησε πρόσφατα το δικαστήριο. Τα παιδιά ζουν στην Ιταλία με τους γονείς που δεν έχουν παντρευτεί ε, και ε, που χωρίζουν και ε, το, ο, πατέρας απαγορεύει εις, την, τη μητέρα να ζήσει με το παιδί πράγμα το οποίο επιτυγχάνει μέσω του δικαστηρίου ε, αλλά τότε ε, ο πατέρας χάνει την επικοινωνία με το παιδί οπότε αν υπάρξει αυτή η διακοπή της επικοινωνίας τι μπορεί να γίνει υπάρχει από τη μία πλευρά η απόφαση του ε, Ιταλικού δικαστηρίου που χορήγησε ένα δικαίωμα επισκέψεως ένα δικαίωμα σαν αυτό που σας περιέγραψα αλλά η μητέρα ε, μερικώς μποϊκοτάρει αυτό το δικαίωμα και εκεί πρέπει να δούμε πώς εφαρμόζονται και εκτελούνται οι αποφάσεις ε, επικοινωνίας. Τι δυνατότητες έχει ο άλλος ο γονιός ο οποίος ζει σε μια άλλη χώρα να ε, εκτελέσει γρήγορα και αποτελεσματικά το δικαίωμα επικοινωνίας και επίσκεψης. Οπότε θα πρέπει να υπάρξουν πιο αποτελεσματικά αποτελεσματικές διεθνείς διαμεσολαβήσεις για να αποφύγουν την αποξένωση και την ρήξη των επαφών διότι πολλές φορές δεν υπάρχουν αρκετές ε, δυνατότητες παρακολουθήσεως ιδίως από το εξωτερικό των περιπτώσεων αυτών. Και καταρχήν απερίφθη η επιστροφή του παιδιού αλλά στη συνέχεια διετάχθη το παιδί να χρειαστεί να επιστραφεί στην Ιταλία και μετά την επιστροφή του παιδιού και μετά από διευκρίνηση του θέματος από τα Ιταλικά δικαστήρια για το ποιος θα πρέπει να έχει την επιμέλεια του παιδιού στο μέλλον τίθεται το νέο ερώτημα πώς γίνεται ε, η επίσκεψη από τον άλλον γονιό. Δηλαδή πώς θα υπάρχει η επαφή και η επίσκεψη με τον άλλο γονιό ο οποίος ενδεχομένως θα ζει σε μια διαφορετική χώρα και δεν θα έχει εύκολη επικοινωνία. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η διατήρηση της επαφής και με τον άλλο γονιό σε διασυνοριακές σχέσεις μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα από την εκτέλεση του δικαιώματος επαφής και επίσκεψης στο εθνικό δίκαιο. Θα πρέπει όμως να έχει ε, ε, προτεραιότητα η επικοινωνία αυτή και αυτό ε, ήδη θεωρείται ότι είναι ένα θεμελιώδης δικαίωμα του παιδιού να έχει επικοινωνία και με τους δύο γονιούς. Νομίζω λοιπόν ότι θα χρειαστούν νέα μέσα διεθνούς διαμεσολάβησης, οικονομική στήριξη για τα έξοδα ταξιδίου και δυνατότητες συνοδευόμενης επαφής. Σας ευχαριστώ για την την προσοχή σας. Ευχαριστώ για αυτά τα σχόλια σε ένα πάρα πολύ δύσκολο το οποίο ποτέ δεν θα λυθεί επαρκώς. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μία διαταγή επικοινωνίας ευρωπαϊκή άμεσα εκτελεστή αλλά η οποία παρόλα αυτά δεν εκτελείται σωστά. Και τώρα ερχόμαστε στο θέμα της απαγωγής των παιδιών σύμφωνα με τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α και εδώ έχουμε ε, δύο μιλήτριες, την ε, κυρία Χίρς καταρχήν. Τζουλιάνα Χίρς. Ευχαριστώ πολύ. Μιλώ εκ μέρου ε, του αναπληρωτή γενικού γραμματέα μας του William Duncan, ο οποίο δυστυχώ δεν μπόρεσε να παραστεί σημερινή συνεδρίαση. Οπότε θα εκφωνήσω το λόγο του εκ μέρους του. Θα μιλήσω για την ε, παράνομη απαγωγή των ε, παιδιών και την ε, σχέση με, τον, με τις Βρυξέλλες 2α. Η Σύμβαση της Χάγης έχει σήμερα 82 συμβαλόμενα μέρη, κράτη-μέλη, και για την ώρα αποτελεί το βασικό εργαλείο που εξασφαλίζει την γρήγορη επιστροφή των απαχθέντων παιδιών ε, μεταξύ των ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το γεγονός βέβαια ότι η λειτουργία ε, της σύμβασης έχει συμπληρωθεί από τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α. Γι' αυτό το λόγο το αποτέλεσμα αυτής της συμπλήρωσης που δείχνει ακριβώς πόσο μεγάλο επίπεδο ολοκλήρωσης μπορεί να υπάρχει σε περιφερειακό επίπεδο, σκοπό είχε καταρχάς ε, να μειώσει τις ε, προθεσμίες των διαφόρων διαδικασιών, δηλαδή μικρότερες χρονικές προθεσμίες σε σχέση με τις ε, δικαστικές διαδικασίες που προβλέπονται από τη Σύμβαση της Χάγης, όπως επίσης και να ενισχύσει τις αρχές των χωρών από τις οποίες οποίε έχουν απαχθεί τα παιδιά. Ο αριθμό των συμβαλωμένων μερών ε, της σύμβασης αυξάνεται συνεχώς και η τελευταία χώρα που ε, προσχώρησε ήταν το Μαρόκο, η πρώτη αραβική χώρα της ευρωμεσογειακής περιοχής ε, και Κάποια κράτη-μέλη επίσης προετοιμάζουν την προσχώρησή τους, όπως η Ρωσία, η Σιγκαπούρη, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Κένια και οι Φιλιππίνες. Μία από τις μεγάλες προκλήσεις ε, όσον αφορά την αντιμετώπιση του διεθνούς ε, προβλήματος ε, της απαγωγής των παιδιών είναι η εξέβρεση μιας εγκεκριμένης βάσης συνεργασίας με κράτη από τον Ισλαμικό κόσμο. Είναι γνωστό ότι ο αριθμός των απαγωγών από ευρωπαϊκές χώρες σε χώρες όπως η Αίγυπτος, η Λιβύη, το Πακιστάν ή κάποιες από τις χώρες Περσικού κόλπου αυξάνονται συνεχώς. Οι προσπάθειες βελτίωσης συνεργασίας έχουν συμπεριλάβει διεθνείς συμφωνίες, όλο και μεγαλύτερη χρήση διαμεσολάβησης, όπως αναφέρεται για παράδειγμα, ε, αναφέρεται και ήδη σε πολλούς λόγους σήμερα που ακούστηκαν σήμερα, όπως και προσπάθειες ε, εναντίον ενός ε, φαινομένου που έχει πολλές φορές ε, αναφερθεί σήμερα και που σκοπό έχει την καλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ των νομικών συστημάτων των εμπλεκομένων χωρών, όπως για παράδειγμα η διαδικασία της Μάλτας που ξεκίνησε στο πλαίσιο της Σύμβασης της Χάγης πριν από πέντε χρόνια με σκοπό την προώθηση διαλόγου μεταξύ των δικαστών ε, των κρατών μελών ε, που ε, έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσει κανείς ότι η βελτιωμένη συνεργασία έχει μια ε, στέρεα νομική βάση όπως αυτή που προβλέπει η Σύμβαση της Χάγης του 1980. Είναι σημαντικό να διερευνήσει κανείς εναλλακτικές επιλογές όπως η διαμεσολάβηση και επίσης ε, υπάρχει και μια πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της διάσκεψης της Χάγης, ε, στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μάλτας που ενθαρρύνει την ανάπτυξη των δομών διαμεσολάβησης σε χώρες που δεν συμμετέχουν στη Σύμβαση της Χάγης που είναι βέβαια πολύ επικοδομητική και για τη διαμεσολάβηση των χωρών που, ε, μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν ε, στη Σύμβαση της Χάγης. Όμως ε, είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να παραμείνει κάτι τέτοιο χωρίς νομικό πλαίσιο. Δεν επαρκεί αυτό γιατί υπάρχει περίπτωση σε αυτές τις περιπτώσεις απαγωγών παιδιών ο γονέας που κάνει την απαγωγή τελικά να ε, ευνοηθεί και ο άλλος γονέας ε, να προσπαθεί απλώς τελικά να διαπραγματευτεί τα δικαιώματα επικοινωνίας με το παιδί του. Οπότε χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο για την υποστήριξη της διαμεσολάβησης σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Επίσης ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αν υπάρχουν και συμφωνίες πρέπει να γίνονται αποδεκτές στα διάφορα νομικά συστήματα και επίσης αν δεν υπάρχουν συμφωνίες πρέπει να βρεθεί μια δικαστική λύση για τις περιπτώσεις αυτές. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε περισσότερες εξελίξεις στον τομέα αυτό. Πρώτον, συνεχίζοντας την προσπάθεια οικοδόμησης εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ των νομικών συστημάτων μέσω διαδικασιών όπως η διαδικασία της Μάλτας και του προγράμματος ε, του Ευρωμεσογειακού, όπως επίσης και ε, δίνοντας μεγαλύτερες ευκαιρίες ε, συνεργασίας μεταξύ δικαστών και αξιωματούχων των ε, διαφόρων χωρών. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο διασκέψεις που έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο της διάσκεψης της Χάγης, ε, μία στο Μαρόκο, σε συνεργασία με το πρόγραμμα ε, το ευρωπαϊκό ΤΑΙΒΕΞ για το Δεκέμβριο του 2010 και μία ακόμη στο Κατάρ τον Απρίλιο του 2011. Οπότε βέβαια η διάσκεψη της Χάγης συνεχίζει τις προσπάθειές της ε, για την βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ε, κρατών μέσω περιφερειακών διασκέψεων. Ένα δεύτερο σημείο που είναι επίσης σημαντικό και το οποίο πρέπει να το σημειώνει κανείς όταν μιλά για την ανάπτυξη μεγαλύτερων προσπαθειών στον τομέα αυτό είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να τονίζουμε τις κοινέ αξίε. Ε, που αναφέρονται στο πλαίσιο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Παιδιών του ΟΗΕ. Γιατί είναι μια βασική, είναι μια βάση ε, για να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη και ε, ο σεβασμός. Όλα τα κράτη-μέλη συμφωνούν ότι το παιδί έχει θεμελιώδες δικαίωμα να διατηρεί τακτικές επαφές και προσωπικές σχέσεις με τους δύο του γονείς. Και επίσης ε, η σύμβαση του ΟΗΕ στο άρθρο 11 αναφέρεται και στο, στην υποχρέωση του κράτους να συνεργαστεί με σκοπό την ε, ε, καταπολέμηση της παράνομης απαγωγής και της μη επιστροφής του παιδιού. Οπότε αν αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα θα μπορέσουμε να λύσουμε πιο αποτελεσματικά το πρόβλημα στο μέλλον. Ε, για πάνω από 25 χρόνια υπάρχει η Σύμβαση της Χάγης και βεβαίως αντιμετωπίζει και πολλές προκλήσεις. Και θα ήθελα να σας αναφέρω εννέα από τις προκλήσεις αυτές. Η πρώτη είναι Πώ είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε ότι οι διαδικασίε τη σύμβαση λειτουργούν σωστά και ότι ε, η επιβολή γίνεται και με ευαισθησία και με αποτελεσματικότητα. Πώ να εξασφαλίσουμε σε περιπτώσει οικογενειακή βία, για παράδειγμα, ότι το άρθρο 13 και οι σχετικέ παρεκκλήσει εφαρμόζονται σωστά και ότι η επιστροφή του παιδιού γίνεται ε, υπό συνθήκε ασφαλείας τόσο για το παιδί όσο και για τον γονέα που το συνοδεύει. Τρίτον, πώ να διατηρήσουμε διεθνή συνέπεια στην ερμηνεία των βασικών αρχών του εργαλείου αυτού. Τέταρτον, πώ να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των κεντρικών αρχών, ώστε να είναι ομαλή ε, αποτελεσματική και γρήγορη, πώς να, πώς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αποτελεσματικής πρόσβασης σε διαδικασίες από τη μία σε σχέση και με τον γονέα που κάνει την απαγωγή αλλά και με τον γονέα που μένει πίσω ε, και επίσης σε σχέση με την αποτελεσματική ε, διαδικασία στις χώρες, στη χώρα της απαγωγής και στη χώρα στην οποία πρέπει να επιστραφεί το παιδί. Έκτον, πώς να ενθαρρύνουμε την ευαισθητοποίηση αλλά και την εφαρμογή των προληπτικών στρατηγικών συμπεριλαμβανομένης μια εγκεκριμένη προσέγγισης για το θέμα της οικογενειακής επανεγκατάστασης. Έβδομον, πώς να βελτιώσουμε την υποστήριξη διασυνοριακών δικαιωμάτων επαφών μεταξύ γονέων και παιδιών, κάτι το οποίο έχει ήδη συζητηθεί. Και οχτώ, ε, πώς να εξασφαλίσουμε ότι οι δικαστές ε, στα 82 συμβαλώμενα μέρη της σύμβασης ε, είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν ε, τα προβλήματα τέτοιων υποθέσεων ε, ε, και ότι μέσω δικτύωσης και άμεσης δικαστικής επικοινωνίας έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν την απαραίτητη αμοιβαία εμπιστοσύνη ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και σε άμεση να συμμετέχουν σε άμεση επικοινωνία για την επίλυση των διαφόρων υποθέσεων. Τελευταία, ε, τελευταίο σημείο που θα ήθελα να θέσω είναι πώς θα υπάρχει μια νοοτροπία διαπραγμάτευσης και συμφωνίας ε, γύρω από τα ζητήματα αυτά και πώς να χρησιμοποιηθεί η διαμεσολάβηση και άλλα είδη ε, επίλυσης διαφορών όταν έχουν γίνει απαγωγές. Αυτές είναι μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η λειτουργία της Σύμβασης της Χάγης Βέβαια, ελπίζει ότι με την ε, υποστήριξη των ε, ε, εταίρων της σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο να μπορέσει να τα επιλύσει. Για παράδειγμα, ανάπτυξη εγχειριδίων καλής πρακτικής. Έχουμε ελάχιστους ε, τέτοιου είδους ε, ε, οδηγούς, όπως για παράδειγμα κάποιους που αφορούν την επιβολή, την πρόληψη, την επικοινωνία γονέα με το παιδί και για τη διαμεσολάβηση. Θα σας πω ορισμένα πράγματα γι' αυτό σε λιγάκι. Ένα δεύτερο μέτρο είναι η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών μέσω του Ινκαντάτ, για παράδειγμα που είναι η βάση δεδομένων ε, απαγωγών παιδιών, όπου αναφέρονται οι διάφορε εθνικέ αποφάσει σε διάφορε γλώσσε, συλλογή στατιστικών πληροφοριών ε, σε σχέση με την ε, λειτουργία τη σύμβαση, κάτι ακόμη, ανάπτυξη του, δικαστικού, του Διεθνού Δικαστικού Δικτύου τη Χάγη, στο οποίο σήμερα συμμετέχουν 50 δικαστές. Επίσης, τακτικές αναθεωρήσεις της σύμβασης μέσω ειδικών επιτροπών επιτροπών που θα συνεδριάζουν. Η επόμενη μάλιστα θα λάβει χώρα τον Ιούνιο του 2011 και βέβαια κάτι το οποίο είναι επίση πολύ ενδιαφέρον. Είμαστε σε αρκετά πρώιμο στάδιο συζήτησης για το κατά πόσο θα έπρεπε να συμπληρωθεί με πρωτόκολλο η σύμβαση ε, με κάποια από τα μέτρα. Βλέπω ότι δεν έχω πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, ούτως ή άλλως έχετε και την ε, παρουσίασή μου στο φάκελό σας. Θα ήθελα απλώς να ε, αναφερθώ στο ότι έχουμε δύο οι πρωτοβουλίες, τον οδηγό και το ε, πρόγραμμα το οποίο ανέφερα και θα ήθελα να πω ότι το πρόβλημα της διεθνούς απαγωγής παραμένει για μας ε, ένα σημαντικό πρόβλημα. Η διεθνής κινητικότητα έχει αυξηθεί και μπορεί να δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στο παιδί όταν οι γονείς τους δεν έχουν πια την σχέση που είχαν στο παρελθόν και και είναι ο καλύτερο τρόπο η σύμβασή μα να μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα τη μη επιτροφή των παιδιών. Η σύμβαση αυτή ε, σκοπό έχει να καταβάλει ακόμη περισσότερες προσπάθειες ώστε να παραμείνει λειτουργική, αποτελεσματική και για να προστατεύσει ε, τα παιδιά όσο το δυνατόν περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ε, τώρα η κυρία Χριστίνα Μπλακ Λαός, η οποία είναι νομικός από την Law Society της Αγγλίας και της Ουαλίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Α, αντίθετα με την συμπατριώτησά μου σήμερα το πρωί σας διαβεβαιώ ότι δεν είμαι κλασική Αγγλίδα. Είμαι η Κριστίνα ε, Μπλάκλος, δικηγόρος στην Αγγλία και στην Ουαλία και προεδρεύω ε, της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Οικογενειακού Δικαίου. Είμαστε υπεύθυνοι για 144.000 δικηγόρους και έχουμε ένα γραφείο και εδώ στις Βρυξέλλες για να εξασφαλίζουμε ότι οι απόψεις του νομικού επαγγέλματος αντιπροσωπεύονται στα όργανα των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προάγουν τη σωστή νομοθεσία και την πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την βοήθεια που μου παρήχαν κατά την προετοιμασία αυτής της εργασίας. Η Τζουλιάνα Χέρς σας μίλησε για την απαγωγή των παιδιών στο πλαίσιο της Σύμβασης της Χάγης. Εγώ θα αναφερθώ στα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α και θα σας κάνω μια γενική επισκόπηση των βασικών διατάξεων. Θα διαφωτίσω επίσης του πώς έχει οικοδομηθεί αυτός ο κανονισμός στο καθεστώς της Χάγης. Επίσης θα σας πω κάποια πράγματα και από τη δική μου δοσηδικία, τη Νέα Αγγλία και την Ουαλία και θα υποδείξω και κάποιους τομείς για μελλοντική εργασία. Καταρχήν, ας πούμε, τι εννοούμε με τον όρο απαγωγή παιδιού. Υπάρχουν δύο μορφές απαγωγής του παιδιού, είτε παράνομη απομάκρυνση, είτε κράτηση. Και οι δύο μορφές πρέπει να παραβιάζουν το δικαίωμα γονική επιμέλεια, σύμφωνα με τον νόμο του κράτου μέλους, όπου το παιδί έχει τη συνήθεια διαμονή του, αμέσως πριν από την απομάκρυνση ή την κράτησή του. Όπω με όλου του τομεί του οικογενειακού δικαίου, οι περιπτώσει αυτέ ε, είναι επιτακτικέ συγκινησιακές και αγγίζουν την χαρτιά, τον πυρήνα της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων. Για το λόγο αυτό η νομοθεσία στους τομείς αυτούς ε, περιέχει κανόνες ε, για τη σωστή αντιμετώπιση και οι κεντρικές αρχές σε κάθε χώρα ε, συνεργάζονται ταχύτατα μεταξύ τους για να προστατεύσουν τα δικαιώματα του παιδιού. Ο κανονισμός Βρυξέλλες 2α στόχο έχει να διασφαλίσει πραγματικά την άμεση επιστροφή του παιδιού. Ενθαρρύνει ε, ταχύτατη και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Ο κανονισμός ορίζει πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα για τις περιπτώσεις αυτές και η προσοχή εστιάζεται στη διεξαγωγή των διαδικασιών με τους ταχύτατους δυνατούς ρυθμούς σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και εν πάση περιπτώσει εντός του χρονοδιογράμματος των έξι εβδομάδων. Η ανάγκη για ταχύτητα ε, αντικατροπτίζεται και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όταν υλοποιεί και ε, δημοσιεύει αποφάσεις για προκατακτικά ζητήματα. Ε, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε αυτή η διαδικασία για την απαγωγή παιδιών πάρα πολύ αποτελεσματικά. Ο κανονισμός επίσης επιταχύνει και απλοποιεί τις διαδικασίες επιβολής του νόμου. Ο κανονισμός παρέχει ε, την άμεση αναγνώριση και εφαρμογή των αποφάσεων σε άλλα κράτη-μέλη χωρίς περαιτέρω ανάγκες καταγραφής ή αναγνώρισης ή διακήρυξης της εκτελεστότητας και παρέχει ένα σχετικό πιστοποιητικό. Ο γενικό κανόνα είναι ο εξή. Όταν απάγεται ένα παιδί από ένα κράτο μέλο σε ένα άλλο κράτο μέλο, το δικαστήριο όπου το παιδί είχε τη συνήθεια διαμονή του αμέσω πριν από την απαγωγή του, το κράτο χώρου του κράτου μέλου τη προέλευση, εξακολουθεί να έχει την αρμοδιότητα. Παρόλο που το παιδί τώρα διαμένει σε άλλη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το δεύτερο κράτο μέλο, το μέλο τη αίτηση, έχει αρμοδιότητα μόνο σε δύο πολύ συγκεκριμένε περιπτώσει περιπτώσεις. Όταν το παιδί έχει αποκτήσει συνήθη διαμονή στην χώρα και το, η γονική επιμέλεια ε, έχει συνενέσει στην απαγωγή ή όταν το παιδί έχει συνήθη διαμονή και έχει παραμείνει τουλάχιστον επί ένα χρόνο στο νέο κράτος μέλος. Η συνήθις ε, διαμονή είναι αποφασιστική σημασίας, αλλά δεν υπάρχει ορισμός στον κανονισμό και αυτό εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια. Μια καινοτομία στον κανονισμό Βρυξέλλες 2α σε σχέση με τη Σύμβαση της Χάγης είναι ότι ε, θέτει τα συμφέροντα του παιδιού στην καρδιά της διαδικασίας. Αυτό ε, σημαίνει ότι το δικαστήριο ακούει το παιδί. Υπάρχει μια διαδικασία ακρόασης. Αυτή δεν ορίζεται από τον ίδιο τον κανονισμό και εναπόκειται και πάλι ε, στα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν αυτό το μηχανισμό ακρόασης. Μερικά λόγια τώρα για την δική μου δοσηδικία. Σύμφωνα σύμφωνα με την νομοθεσία του 1984 αποτελεί ποινικό αδίκημα να αφαιρείται ένα παιδί από το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς τη συνένεση του παιδιού που έχει τη γονική ευθύνη για αυτό το παιδί. Η κεντρική αρχή στην Αγγλία και την Ουαλία είναι ο καγκελάριος του νόμου, ο, ο οποίος είναι υπεύθυνο είναι το σημείο επαφής για τις περιπτώσεις απαγωγής των παιδιών σημειώνεται ότι υπάρχουν τρία επίπεδα αρμοδιότητας αγγλία και ουαλία ε, Σκοτία και Βόρεια Ιρλανδία. Ε, κάθε μία από αυτές έχει διαφορετικά νομικά συστήματα και ούτε ε, η Χάγη ούτε οι Βρυξέλλες 2α μπορούν να υπησέλθουν. Ωστόσο, κάποιες περιπτώσεις μπορούν να παραπεμφθούν. Η Σκοτία και η Βόρεια Ιρλανδία και οι δύο έχουν τις δικές τους κεντρικές αρχές. Δεν επίσης δεν επιβάλλεται κανένα είδος τέλους ή φόρου για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Όταν ένα παιδί λοιπόν έχει απαχθεί στην Αγγλία και στην Ουαλία ή διακρατείται εκεί, οι γονείς κάνουν μια αίτηση για την επιστροφή του παιδιού στη δική τους κεντρική αρχή, του δικού τους κράτους μέλους. Η κεντρική αρχή διαβιβάζει αυτήν την αίτηση ή έρχεται σε άμεση επαφή ο γονέας Εάν ε, πληρούνται οι προϋποθέσεις, τότε παραπέμπεται σε έναν ειδικό έμπειρο δικηγόρο, ο οποίος είναι ενήμερος για τα σχετικά περιστατικά, που έχει εμπειρία. Όλες οι υποθέσεις ακούγονται στο Λονδίνο από το Ανώτατο Δικαστήριο και από το Πρωτοδικείο, συγγνώμη, και διασφαλίζεται η ταχύτατη εκδίκαση των υποθέσεων αυτών. Για παράδειγμα, 21 μέρες είναι το ανώτατο όριο. Το δικαστήριο λοιπόν να ασκεί έλεγχο. Εάν αντιστραφεί η κατάσταση και ένα παιδί απαχθεί σε χώρα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, η υπόθεση παραπέμπεται στο ΑΙΚΑΚΟΥΝ και εκεί αναλαμβάνει κάποιος και πάλι έμπειρος δικηγόρος, ο οποίος συμπληρώνει τις αιτήσει και αναλαμβάνει τη διαδικασία επιστροφής του παιδιού. Η αίτηση και τα σχετικά έγγραφα και τυχόν μεταφράσεις αποστέλλονται στην κεντρική αρχή της χώρας του παιδιού όπου το παιδί κρατείται ή έχει απαχθεί. Παρακολουθείτε λοιπόν η πρόοδος της υπόθεσης, παρέχονται συμβουλές για το αγγλικό δίκαιο και γίνονται όλα όσα, όσα απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η εκδίκαση του περιστατικού. Εν κατακλείδη λοιπόν ο κανονισμός Βρυξέλλες 2α έχει πραγματικά βελτιώσει διαδικαστικά τις ε, περιπτώσεις αυτές συμπληρώνοντας τις ρυθμίσεις ε, της συνθήκης της Χάγης. Οι κύριες καινοτομίες είναι οι αυστηρές προθεσμίες, οι αρχές τοποθέτησης του συμφέροντος του παιδιού στο επίκεντρο της διαδικασίας των αποφάσεων, οι ειδικέ διατάξεις για την ακρόαση του παιδιού ελαχιστοποίηση των λόγων απόρριψης της αίτησης επιστροφής. Ένας γονέας δεν μπορεί να αρνηθεί να επιστρέψει το παιδί, με εξαίρεση την περίπτωση που το άτομο που ζητεί την επιστροφή του παιδιού μπορεί να ακουστεί το ίδιο. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορείτε να δείτε την ομιλία μου για κάποια παραδείγματα, δείχνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα και θα ήθελα να τονίσω τρεις τομείς από το για το 2012 όταν θα αναθεωρηθεί ο κανονισμός. Πρώτον, η έλλειψη ορισμού για την συνήθη διαμονή. Δεύτερον, το ζήτημα για το ποιος έχει το δικαίωμα της επιμέλειας. Είτε και αν ο ορισμός συμπεριλαμβάνει τους ε, άγαμους πατέρες. Και δεύτερον, ο προσδιορισμός της αρμοδιότητας. Θα έλεγα ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και στα τρία αυτά ζητήματα. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω και μια τελική σύσταση. Την εξής ε, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο κατάρτισης για όλους τους νομικούς, για όλα τα νομικά επαγγέλματα που εμπλέκονται. Και αυτό είναι προϋπόθεση για τη γρήγορη και ορθή εφαρμογή του κανονισμού θεωρώ ότι τα θέματα αυτά πρέπει να εξετασθούν και μέσω των διάβλων χρηματοδότησης της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και για την παραπομπή εις ε, την κατάσταση στην ε, πόλη σας ε, ε, θέματα τα οποία πραγματεύονται πολλοί κανονισμοί θα μπορούσαμε ίσως να συμφωνήσουμε εμείς σε έναν ορισμό και να τον αφήσουμε στη διάκριση των κρατών μελών. Τώρα ερχόμαστε στο θέμα των παιδιών στις δικαστικές διαδικασίες και καταρχήν ε, την ε, συμμετοχή του παιδιού στις ακροματικές διαδικασίες και δίνω το λόγο στην κυρία μία ε, ράη. Ευχαριστώ όπως και ο προηγούμενος ε, ομιλητής ε, είμαι δικηγόρος στη Σουηδία και μου ζήτησαν να εξετάξω τα, την προστασία των παιδιών στις ε, ακροαματικές διαδικασίες στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα καταρχήν να πω ορισμένα πράγματα για την ε, Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την εξάσκηση των δικαιωμάτων του παιδιού που ε, συμφωνήθηκε στο Στρασβούργο 25 Ιανουαρίου 1996. Γι' αυτό τα παιδιά πρέπει να έχουν πληροφόρηση για να μπορέσουν να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους. Επίσης τονίστηκε ότι τα παιδιά ε, θα πρέπει ε, να ε, έχουν υπόψη τους το σημαντικό ρόλο των γονέων για την προστασία και πρόθεση των δικαιωμάτων τους και τα παιδιά πρέπει να επιτηρούν όπως άλλωστε και τα κράτη-μέλη την παρακολούθηση αυτή και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία προηγουμένως μιλήσαμε για διαμεσολάβηση. Πρέπει να σας πω ότι στη Σουηδία υπάρχει ένα ε, ε, Ινστιτούτο που λέγεται ε, συνεργατικές συζητήσεις όπου υπάρχουν εξοδικαστικές διαδικασίες οι οποίες μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνίες. Ε, όπως ξέρετε ο κανονισμός Βρυξέλλες 2 έχει επεκτείνει ε, αυτές τις διατάξεις και αναφέρεται και στις επιθυμίες του παιδιού το οποίο απετέλεσε μία σημαντική αλλαγή σε σχέση με ε, τον κανονισμό Βρυξέλλες 2. Αν αναφερθώ και συγκρίνω την κατάσταση στα κράτη-μέλη και στην νομοθεσία τους, πρέπει να πω ότι τα παιδιά προστατεύονται, εισακούονται, αλλά υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των διατάξεων βάσει των οποίων εφαρμόζονται τα δικαιώματα και λαμβάνονται υπόψη. Έχουν υπάρξει ορισμένες ε, ε, ε, αλλαγές, ιδίως όσον αφορά αφορά τη συμμετοχή των παιδιών στις ακροαματικές διαδικασίες το πώς ε, εκπροσωπούνται τα παιδιά, πώς ε, λαμβάνονται υπόψη οι απόψει τους. Αλλά σε όλους αυτούς τους τομείς ακόμη πολλά μένουν ακόμη να γίνουν, διότι ε, όλα τα κράτη-μέλη θέλουν να προστατεύσουν τα δικαιώματα των παιδιών ή στις ακροματικές διαδικασίες, αλλά υπάρχουν διαφορές. Και οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες ώστε θα έπρεπε να εξεταστούν εκ του και θα επανέλθω στο σημείο αυτό. Είμαστε πιο συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για το πόσο θα εισακούονται τα παιδιά στις ακροματικές διαδικασίες και ε, να ε, υπάρξουν περισσότερες ε, ενεργές συμμετοχές των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Στα περισσότερα κράτη τα παιδιά μπορούν να παριαστούν σαν μάρτυρες στις αστικές διαδικασίες αλλά σε πολλές άλλες τα δικαστήρια διστάζουν να ακούσουν τα παιδιά σε ορισμένες χώρες ε, δεν μπορούν να συμμετάσχουν καθόλου στις δικαστικές διαδικασίες, σε άλλα από μία ηλικία και μετά. Ε, ε, πρόκειται όμως για θέματα που τους αφορούν, όπως είναι η επιμέλεια, η κυδαιμονία, άρα θα έπρεπε και οι δικές τους απόψεις να ληφθούν υπόψη. Το πώς αυτό θα επιτευχθεί είναι θέμα διαφορετικής αντιμετωπίσεως στα διάφορα κράτη και γι' αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να δούμε πιο κοντά. Ε, όπως είπα μπορούν να υπάρξουν και διαφορετικοί τρόποι μέσω των γονέων, μέσω των κοινωνικών λειτουργών, μέσω εμπειρογνωμόνων. Ε, ε, οι τρίτοι αυτή συνήθως καθορίζονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες και δεν είναι εξίσου σημαντική ίσως αλλά έχουν κάποια σημασία. Επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν τα παιδιά με το δικαστήριο μέσω παιδοψυχολόγων ή άλλων ειδικών. Το δικαστήριο μπορεί να ακούσει το παιδί είτε μόνο του ή μαζί με τον ψυχολόγο του οπότε ίσως μπορεί να ε, ε, εισακουστεί και ε, σε πολύ νεαρή ηλικία δηλαδή ήδη από 7 ή 8 ετών σπανίως το παιδί εκπροσωπείται χωριστά. Πράγμα όμως το οποίο είναι μειονέκτημα και θα έπρεπε να διορθωθεί. Όταν ένα παιδί συμμετέχει στη διαδικασία σύμφωνα με το στις Βρυξέλλες 2 2B εκπροσωπείται είτε από τον ειδικό ο παιδοψυχολόγο ή από τους γονείς του. Θα πρέπει όμως να υπάρξει σοβαρή Υπάρχει παρακολούθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και γι' αυτό μια χώρα σκοπεύει μάλιστα να κάνει δημοψήφισμα επί του θέματος για να ε, βελτιώσει την προστασία του παιδιού όσον αφορά την κυδαιμονία, την επιμέλεια, την ε, πρόσβαση και επικοινωνία με το παιδί και ούτω καθεξής. Το παιδί έχει διάφορα δικαιώματα και ε, θα πρέπει ίσως να υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση. Η Σουηδία έχει αναγνωρίσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την εξάσκηση των δικαιωμάτων του παιδιού και έχει κάνει ορισμένες παρατηρήσεις σε τμήματα της νομοθεσίας. Προβλέπετε ότι σύντομα θα υπάρξει ε, μία πρόταση να συμπεριληφθεί αυτή η σύμβαση εις την Σουηδική νομοθεσία για να ενισχύσει τα δικαιώματα του παιδιού στην Σουηδία και όπως είπα υπάρχει η δυνατότητα για το παιδί να ε, εκφραστεί σχετικά με την προτίμησή του σχετικά με το, την ε, διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί αλλά πολλές φορές η εκπροσώπηση και συμμετοχή σε δικαστικές διαδικασίες διαφέρει και καμιά φορά το παιδί δεν συμμετέχει καθόλου. Μία μελέτη στην Αγγλία είπαν ε, οι μας λέει ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι το παιδί δεν πρέπει να μπλέκεται καθόλου. Και επίσης στη Γερμανία ε, ελέγχθη ότι οι περισσότεροι δικαστές, 88% δεν ήθελαν το παιδί να συμμετέχει καθόλου στη διαδικασία. Και ε, πολλές φορές ε, σε υπάρχουν χώρες όπου το παιδί συμμετέχει μόνο σε 2,5% των περιπτώσεων και σε άλλες χώρες, ακόμη και στη Σουηδία, όπου δεν συμμετέχει καθόλου. Στην πραγματικότητα όμως έχουν δικαίωμα τα παιδιά να έχουν εκπροσώπηση σε 1,6% των περιπτώσεων στη Γερμανία και 10% μπορεί να φτάσουν σε περιπτώσεις ή στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει όμως να εξετάζουμε πιο προσεκτικά τις απόψεις του παιδιού, διότι κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να εξετάσουμε συγκεκριμένη συγκεκριμένα το, τα μέσα με τα οποία θα πρέπει να ε, ακούμε τα παιδιά, ε, πώς δηλαδή θα πρέπει να συμμετέχουν στις ε, διαδικασίες. Προηγουμένως αναφέρθηκα ή στους μεσολαβητές οι οποίοι είναι χρήσιμοι, αλλά κάθε χώρα χρειάζεται να εκπαιδευτεί και να έχει κατευθυντήριες γραμμές διαφορετικά μεταξύ χωρών οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες μεγάλες και μεταξύ των παιδιών τα οποία υπάρχουν στις χώρες αυτές υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Έχω εξετάσει το θέμα των ορισμών που ήδη αναφέρθηκε ότι χρειαζόμαστε πιο συγκεκριμένους ορισμούς όσον αφορά το συνήθι τόπο διαμονής, ε, την επιμέλεια και άλλα θέματα ε, αλλά πιστεύω στα διάφορα κράτη εννοούμε διαφορετικά πράγματα χρησιμοποιώντας τους ίδιους όρους άρα υπάρχει επίγουσα ανάγκη για κατάρτιση ορισμών επίσης. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτή ήταν μία καλή πρόταση ε, να διατυπώσει κάποια χώρα προτάσεις για το πώς θα εισακούονται τα παιδιά και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα που ε, είναι η αναγνώριση της ε, ευθύνη, γονικής ευθύνης βιολογική γονής έναντι νομίμων γονιών και αμοιβαία αναγνώριση των ε, συμφωνιών ε, βιολογικών γονέων. Ε, επ' αυτού του θέματος θα μας μιλήσει η κυρία Βελίνα Τοντόροβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η παρουσίασή μου σκοπό έχει να παρουσιάσει το περίπλοκο ζήτημα που έχει να κάνει με το ουσιαστικό οικογενειακό δίκαιο σε σχέση με τις παρένθετες εγκυμοσύνες, όπως επίσης και σε σχέση με τα ζητήματα διεθνούς ιδιωτικού δικαίου που αφορούν το θέμα αυτό θα κάνουμε και προτάσει σε σχέση με το πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Είναι γεγονός ότι η αναπαραγωγική ιατρική έχει πάρα πολύ βελτιωθεί, όπω επίση, επειδή υπάρχουν και διάφορε μορφέ οικογένεια πλέον και υπάρχει και το θέμα τη αναγνώριση των δικαιωμάτων των παιδιών, έχουν, έχει επηρεαστεί η όρο τη ε, της του γονέα. Μέχρι τώρα ε, ο, ο νόμιμος ήταν ε, αυτό ο οποίο είχε γενετική σχέση με το παιδί. Όμως το γεγονός ότι υπάρχουν πλέον ε, δωρεές ε, και νέες τεχνολογικές εξελίξεις είναι γεγονός ε, ότι μερικές φορές η ιδιότητα του γονέα δεν είναι υποχρεωτικά αυτή του βιολογικού γονέα. Σήμερα μπορούν να γεννιούνται μωρά που δεν έχουν κανένα, καμία γενοτική σχέση με τους γονείς τους ε, ή μερικές φορές αποτέλεσμα συμβατικών ε, ε, σχέσεων μεταξύ ενηλίκων. Οι παρένθετες εγκυμοσύνες, για παράδειγμα, δημιουργούν πολλά ηθικά διλήμματα τα οποία τα συζητιούνται και σε ακαδημαϊκό επίπεδο αλλά και σε πάρα πολλά έγγραφα πολιτικών. Η παρένθετη εγκυμοσύνη είναι το εξής. Η γυναίκα ε, εγκυμονεί σε παιδί που ε, θα ανήκει σε διαφορετικό άνθρωπο από τη στιγμή της γέννησής του. Αυτό σημαίνει ότι ε, υπάρχουν κάποια νομικά ζητήματα ε, τα οποία είναι πολυάριθμα. Πώς μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι ισχύει η ιδιότητα του γονέα ε, πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε τις ιατρικές πρακτικές, ε, πώς είναι δυνατόν ε, τα, οι γονείς που προβαίνουν σε αυτή τη λύση να ληφθούν υπόψη σε ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και υπάρχει και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Υπάρχει το θέμα της διασυνοριακής παρένθετης μητρότητας που δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα σε σχέση με το νομικό καθεστώς του παιδιού και σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού και την ταυτότητα του παιδιού οι νομοθεσίε των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό διαφορετικά. Μόνο δύο εκφράζουν ε, νομοθεσία ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα και η Ελλάδα όμως είναι διαφορετική πρακτική που ισχύει. Ε, κάποια κράτη-μέλη δέχονται την πρακτική και κάποια άλλα κράτη-μέλη δεν δέχονται καθόλου αυτήν την ε, πρακτική. Ε, υπήρχαν ε, κάποιοι περιορισμοί σε επίπεδο εθνικής ε, νομοθεσίας ε, για τα θέματα της παρένθετης εγκυμοσύνης, ένα θέμα στο οποίο ενέσκυψαν πάρα πολλοί ακαδημαϊκοί. Συχνά η νομική ιδιότητα του γονέα δεν προκύπτει αμέσω από τη Συμφωνία Παρένθετης μητρότητα. Οι προβλεπόμενοι γονείς ε, δεν έχουν ιδιότητα του γονέα μόνο και μόνο λόγω της Συμφωνίας αυτής, ε, ακόμη και αν το παιδί έχει κάποιο βιολογικό σύνδεσμο μαζί του, Αυτό σημαίνει ότι η Συμφωνία από μόνη τη δεν είναι εφαρμοστέα. Και η ιδέα είναι ότι η παρένθετη μητέρα η οποία σε κάθε κράτο μέλο, εκτό από την Ελλάδα, θεωρείται η νόμιμη μητέρα του παιδιού, που ε, δεδομένου του ότι εκείνη φέρνει στον κόσμο το παιδί, δεν δεσμεύεται όμως με κανέναν συμβατικό, συμβατική υποχρέωση να παραδώσει το παιδί της. Δεν είναι υποχρεωμένη να παραδώσει το παιδί στους προβλεπόμενους γονείς, γονείς που θέλουν να πάρουν το παιδί αυτό, μόνο μόνο νομικά μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα και όχι με τη συγκεκριμένη σύμβαση. Ο σκοπός της Συμφωνίας Παρένθετης Εγκυμοσύνης είναι να βοηθήσει το δικαστήριο να αποφασίσει για τη νομική ιδιότητα του ε, γονέα. Η κρατική νομοθεσία το προβλέπει αυτό είτε μέσω εντολής ε, είτε μέσω υιοθεσία ε, σε σχέση με τους γονείς που προβλέπεται να πάρουν το παιδί γιατί μετά από τέτοιου είδους ε, συμφωνία υπάρχει ληξιαρχική πράξη με το όνομα των, γονικό, των γονέων που προβλέπονται. Μόνο στην ε, Ελλάδα δεν ισχύει αυτό, δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει παρένθετη, συμφωνία παρένθετης εγκυμοσύνης σημαίνει ότι η προβλεπόμενη μητέρα είναι αμέσως η μητέρα του παιδιού. Υπάρχουν απόψεις ότι πρέπει να μην είναι εμπορική πρακτική κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να ρυθμιστεί με κάποιο τρόπο. Και γι' αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μια αρμόδια αρχή. Ε, οι κατοχώρε και, η Βελγία, και για το Βέλγιο ασχολούνται με το ζήτημα αυτό μέσω συγκεκριμένων ηθικών αρχών που έχουν ε, ε, ιδρύσει η ιδέα της ρύθμισης είναι μία πτυχή που καθεστά την παρένθετη μητρότητα πολύ παρόμοια με την υιοθεσία. Το διασυνοριακό, η διασυνοριακή παρένθετη εγκυμοσύνη είναι ένα ε, ζήτημα που είναι αντικείμενο διασυνοριακής αναπαραγωγικής υγείας σε μερικές χώρες. Δεν υπήρχε ε, όμως, δεν υπήρχαν μελέτες για, το θέμα για τα θέματα αυτά. Μόνο προσφάτως ε, εξετάστηκε το θέμα στις ε, πτυχές ε, διεθνούς ιδιωτικού ε, δικαίου. Και κυρίως πρέπει να λυθεί το ζήτημα και λόγω των συνεπειών που έχει για το παιδί από νομικής απόψης, αλλά και για τους ενήλικες. Υπάρχουν σε διασυνοριακό επίπεδο πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, Υπάρχουν ε, ενήλικε στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, το Βέλγιο ε, που έχουν ε, συνάψει συμφωνίες παρένθετη εγκυμοσύνης με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως για παράδειγμα με άτομα στι Ηνωμένε Πολιτείες. Κάποιες χώρε, α πούμε, δεν θεωρούν ότι το ουκρανικό πιστοποιητικό γέννησης ε, είναι ενάντια στην ε, εθνική νομοθεσία, γιατί ακριβώς δίνει την ιδιότητα του γονέα ε, απευθείας στους ενήλικες που έχουν συνάψει τη συμφωνία. Όμω, σε μερικέ περιπτώσεις τέτοιου είδους πιστοποιητικά έχουν κριθεί παράνομα. Μόνο στη Γαλλία υπήρξε μία περίπτωση ε, όπου στο πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού έγραφε απευθεία το όνομα της ε, μητέρας που θα έπαιρνε το παιδί. σε όλες τις περιπτώσεις τα ονόματα των ε, γονέων που θέλουν να λάβουν το παιδί εμφανίζονται στη ληξιαρχική πράξη αλλά μόνο μετά γιατί σε πολλές χώρες η μητέρα που γεννά το παιδί είναι αυτή που θεωρείται νόμιμη μητέρα του παιδού. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ιδιότητα του γονέα τελικά να μην αποδίδεται ε, στον γονέα που έχει στον ενήλικα που έχει συνάψει την ε, συμφωνία με αποτέλεσμα το παιδί να μην έχει κανένα γονιό και να πρέπει να πάει σε κάποιο ε, ίδρυμα. Αυτό συνέβη στη Μεγάλη Βρετανία. Και φυσικά ε, και η ψυχολογική βλάβη που δημιουργείται είναι πάρα πολύ μεγάλη και για τους ενηλίκες και για τα παιδιά. Τώρα, τι είδους ε, ε, δράση μπορούμε να αναλάβουμε. Η νομική ιδιότητα του γονέα, ο νόμιμος γονέας, ε, είναι μια, ένας όρος που είναι ένα ζήτημα οικογενειακού δικαίου. Όμως για την ώρα κανένα από τα διεθνή ε, εργαλεία δεν έχουν απαραίτητες διατάξεις για να μπορέσει να ρυθμιστεί το θέμα αυτό. Και λέγω των διαφόρων, διαφόρων εθνικών νομοθεσιών, είτε από απαγόρευση μέχρι πολύ, πλήρη φιλελε... μέχρι πολύ φιλελεύθερη προσέγγιση παρένθετης ε, μητρότητας, θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό, ένα σύνολο κοινών προδιαγραφών ουσιαστικού δικαίου που ενδεχομένως για την ώρα να μην είναι εφικτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η λύση θα μπορούσε να είναι ένας νέος κανονικό, ε, κανονισμός ε, για την αμοιβαία αναγνώριση τέτοιου είδους συμφωνιών και τον ορισμό του νόμιμου γονέα κατόπιν συμφωνίας παρένθετης μητρότητας ο, γιατί για την ώρα δεν καλύπτεται το θέμα αυτό στο Βρυξέλλες 1 και 2α. Χρειάζονται όμως δύο, δύο στοιχεία. Οι Βρυξέλλες 2α δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που υπάρχει ε, διάσταση απόψεων σε σχέση με το ποιος είναι ο νόμιμος γονέας ε, ένα δεύτερο σημείο που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι η διασυνοριακή παρένθετη μητρότητα είναι ένα πολύ ευρύτερο θέμα ε, που δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό οποιαδήποτε δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν είναι επαρκής ε, για να επιλύσει το πρόβλημα. Μια άλλη λύση θα μπορούσε να είναι να κάνουμε συντονισμένες προσπάθειες ε, σε επίπεδο και Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Σύμβασης της Χάγης για το Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο Πρώτον, για να αντιμετωπίσει, να, εξεταστούν οι διασυνοριακέ πτυχέ του θέματο ε, βάσει συγκεκριμένων υποθέσεων. Και δεύτερον, να υπάρχει μια διεθνή σύμβαση ε, για τι πτυχέ του ιδιωτικού δικαίου τέτοιου είδου ε, συμφωνιών, σύμφωνα με το μοντέλο τη σύμβαση τη Χάγη για τι διασυνοριακέ υιοθεσίε. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να προβλέπουμε καλύτερα τις αποφάσεις προς όφελος των παιδιών και των γονέων, ε, ε, των ενηλίκων που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά και να μην ε, υπάρχουν πρακτικές όπως για παράδειγμα η κατάλευση των γονέων και εμπορία παιδιών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ε, βλέπουμε ότι ε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε και τα δικαιώματα του παιδιών να μην καταλήξουν άπατρίς και οι μητέρες να αναλάβουν όλα τα προβλήματα. Τώρα θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα των διεθνών υιοθεσιών, ποια είναι η ισχύουσα κατάσταση, τι ανάγκη υπάρχει για ε, κοινοτική ενεργοποίηση ε, και αν μπορεί να υπάρξει μία ενιαία ε, πολιτική υιοθεσία και εδώ είχε ασχοληθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η κυρία Ραφαέλα Πρελιάσκο ε, από το Ινστιτούτο ε, για τα Δικαιώματα του Παιδιού στη Φλωρεντία έχει αναλάβει αυτή τη μελέτη και θα μας την παρουσιάσει. Ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε την ευκαιρία καταρχήν να διεξάγουμε τη μελέτη και στη συνέχεια να την παρουσιάσουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Ο κύριος στόχος της ε, μελέτης συνίσταται στην, ε, σε μια συγκριτική ανάλυση των διαφορετικών εθνικών συστημάτων υιοθεσία με στόχο τη δημιουργία ενός σώματος επικαιροποιημένη γνώσης που μπορεί να βοηθήσει στη χάραξη πολιτικής. Λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο που η πολιτική προοπτικές αυτές μπορεί να έχουν στα διάφορα κράτα-μέλη των Ηνωμένων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την τεκμηρίωση από την άλλη πλευρά και από, την, από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά των εθνικών συστημάτων προστασίας του παιδιού. Θα εστιάσω την προσοχή μου κυρίως στις δικαστικές πλευρές, στις πλευρές δικαστικής αρμοδιότητας. Ο στόχος μας ήταν να βρούμε τα ενοποιητικά στοιχεία ε, στην υπάρχουσα νομοθεσία και τα κύρια διακυβεύματα σε σχέση με τις διαδικασίες της υιοθεσία, προσπαθώντας ταυτόχρονα να εντοπίσουμε μείζωνα ρυθμιστικά κανονιστικά ζητήματα και περιπτώσεις σύγκρουσης για τις οποίες πρέπει να προταθούν κοινέ λύσεις. Καταρχήν πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ε, η συγκριτική ανάλυση έγινε μεταξύ των εμπειριών των κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δείχνει πόσο βαθιές αποκλήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν. Οι διαφορές αυτές μπορεί να είναι πολύ οξυμένες τόσο όσον αφορά τα διαδικαστικά θέματα όσο και στη διάρθρωση των ειδικών φορέων. Και όσο αφορά το ρόλο που παίζουν τα δικαστήρια, οι διοικητικές αρχές, οι νομοθετικές αρχές και γενικότερα οι αρμόδιες αρχές. Όσο αφορά συγκεκριμένα τη διαδικασία της υιοθεσίας, και τις ε, συνέπειες της υιοθέτηση αποφάσεων περί υιοθεσίας, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσο αφορά τις διαδικασίες υιοθεσία μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών ή μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών και υπηκών τρίτων χωρών. Σε γενικές γραμμές η υπηκότητα των φετών γονέων δεν αποτελεί προϋπόθεση. Όσο αφορά την εφαρμογή του δικαίου σε συγκεκριμένες χώρες, οι γονείς πρέπει να έχουν απλώς την νόμιμη διαμονή τους σε μια ευρωπαϊκή χώρα η αναγνώριση ξένων αποφάσεων, αλλοδαπών αποφάσεων υιοθεσία είναι αυτόματη μόνο στο πλαίσιο των χωρών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της χάγη. Εάν Ευρωπαίοι πολίτες που διαμένουν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα υιοθετήσουν ένα παιδί μέσω των διαδικασιών της χώρας συνήθως διαμονής, ο ο υιοθετημένος προσλαμβάνει την ίδια υπηκότητα με τους υποψήφιους θετούς γονείς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η χώρα της συνήθους διαμονής τους έχει υπογράψει την ε, Σύμβαση της Χάκης για την Διεθνή Υιοθεσία. Και συνοδεύεται αυτό με ένα πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 23 της εν λόγω σύμβασης. Η εντολή της υιοθεσία πρέπει απλώς να καταχωρηθεί στα ληξιαρχεία έτσι ώστε το παιδί να μπορέσει να αποκτήσει την ίδια υπηκοέτητα ε, όπως αυτή των θετών γονιών του ή του θετού γονέα του. Ε, όσο αφορά τι εντολές ή τι αποφάσεις περί υιοθεσία, αυτές πρέπει να επενδυθούν τη μορφή ε, μια διοικητική πράξης ή μιας δικαστικής απόφασης. Και αυτό είναι απαραίτητο Μάλλον η προϋπόθεση για την ε, αναγνώριση της υιοθεσίας που έχει γίνει αλλού θα πρέπει η διαδικασία της υιοθεσίας ε, να υπηρετεί όλες τις ευρωπαϊκές αρχές της διαδικασίας της υιοθεσίας. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες προβλέπουν ότι όταν γίνεται η υιοθεσία σύμφωνα με νομοθεσία που είναι συμβατή με το εσωτερικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε η εντολή υιοθεσία μπορεί να μην, να μην παράγει τις ίδιες συνέπειες για παράδειγμα, η υιοθεσία μπορεί να μην θεωρείται απλή υιοθεσία, αλλά σύνθετη υιοθεσία. Ε, the Στην έκθεση που ε, τονίζεται ότι η πολλαπλότητα των λύσεων για τη ρύθμιση συγκεκριμένων ζητημάτων δεσμευτικών ημί έχει δημιουργήσει σε μεγάλες εντάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν σκεφτούμε μια πιθανή τροποποίηση του συστήματος στο μέλλον, συστήνουμε την απλοποίηση της διαδικασίας και το συντανισμό των υφιστάμενων συστημάτων, έτσι ώστε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή στρατηγική, η οποία να μην περιορίζεται μόνο στην προσχώρηση ε, της σύμβασης για την υιοθεσία, αλλά που να είναι ανοιχτή η διαδικασία και στα, στα άλλα διεθνή κείμενα που αφορούν τα δικαιώματα των ε, υιοθετημένων παιδιών. Θα άξιζε ε, να είμαστε υπέρ μιας τάσης που ήδη έχει γίνει αποδεκτή, αλλά που μπορεί να ε, εξελιχθεί και περισσότερο μέσω μιας συντονισμένη δράσης για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων όπως την επικύρωση των σχετικών διεθνών συνθήκων, την ε, υιοθέτηση κατάλληλων νομοθετικών μέτρων, μηχανισμών παρακολούθησης, κυβερνητικών προϋποθέσεων, αφιέρωσης πόρων, προαγωγής δραστηριοτήτων και μέτρων για την ε, ευαισθητοποίηση της κοινή γνώμης για τα θέματα της ε, προστασίας των παιδιών και για τα θέματα της υιοθεσία. Ιδιαίτερα όσον αφορά την εντολή υιοθεσία, όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην διαδικασία υιοθεσία, ε, όταν έχουν ευρωπαϊκή υπηκότητα, τότε θα πρέπει να βρίσκονται κοινέ λύσεις και να γίνονται ομόφωνα αποδεκτές οι αποφάσεις περιοθεσίας ε, που έγινε σε ένα ευρωπαϊκό κράτος από όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ε, ανεξάρτητα από το αν μια χώρα έχει προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης ή όχι, αρκεί να έχουν τηρηθεί όλες οι ουσιαστικές προϋποθέσεις. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε προς το παρόν είναι το εξής. Δεν φαίνεται να υπάρχει ανάγκη κωδικοποίησης ε, κάποιων ενιαίων νομικών κανόνων, αλλά ε, σημασία έχει να αναπτύξουμε τα εργαλεία που ήδη έχουμε στη διάθεσή μας και να ε, ελέγξουμε αν και κατά πόσο στην, στο ιδιωτικό δίκαιο οι κανόνες του ιδιωτικού δικαίου μπορούν να επηρεαστούν από τις κανόνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η σύνταξη εγγράφων για τις αρχές του δικαίου περιοθεσίας και συγκεκριμένα του διεθνούς δικαίου περιοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καταφέρει μπορεί να παραπέμπει στις διάφορες ε, εθνικές νομοθεσίες σε σχέση με τα βασικά, τα οποία πρέπει να υπηρετούν όλα τα κράτη-μέλη. Και πρέπει επίσης να γίνει και μια καμπάνια ευαισθητοποίησης. Η απουσία ε, νομοθετικής αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασφαλώς είναι σημαντικός παράγων, αλλά όχι ο πιο σημαντικός. Το πρώτο βήμα θα ήταν να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, να εκπονηθεί ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς. Μια πιο λεπτομερή ανάλυση των θεμάτων θα την βρείτε στην σχετική έκθεση. Μπορείτε να την κατεβάσετε από, την, ε, από τον διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τον δικό μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και για το αποτέλεσμα και για την απαρίθμηση των πολλών κανονισμών με τους οποίους ε, ε, πρέπει να ασχοληθούμε. Και τώρα θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στην αντιπρόεδρό μας κυρία Αντζελίλη για να μπορέσει να μας πει τι, με τι ασχολείται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους διοργανωτές αυτής της ε, σημαντικής ευκαιρίας ε, προβληματισμού. Θα περιοριστώ να παρουσιάσω το καθήκον μου ως διαμεσολαβητή, ως συντονίστριας ευρωπαϊκής. Καταρχήν θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν το πρώτο όργανο της Ένωσης που κατανόησε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων θα οδηγούσε και στην ε, αύξηση του αριθμού των οικογενειών που απαρτίζονται από περισσότερες της μία εθνικότητες ή υπηκότητες με όλα τα καλά και τα προβλήματα που αυτό μπορεί να επιφέρει στην περίπτωση του χωρισμού. Το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο ακριβώς δημιούργησε τη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ήδη το 1986 ε, για τα προβλήματα των οικογενειών αυτών πολύ σημαντικό γιατί την εποχή εκείνη η Ευρωπαϊκή Ένωση ονομαζόταν ακόμα Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και δεν ε, καθόλου δεν συζητούσε ούτε καν κάποια ελάχιστη αρμοδιότητα για την ε, πολιτική συνεργασία και πολύ λιγότερο για το οικογενειακό δίκαιο. Το ζήτημα ήταν και είναι για μια σημαντική πρωτοβουλία γιατί και τώρα που αρχίζουμε να έχουμε στοιχεία βλέπουμε ότι πιστοποιείται η σημασία αυτής της διαμεσολάβησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγους μήνες μας ανέφερε ότι κάθε χρόνο στην Ευρώπη ε, ε, πραγματοποιούνται 300.000 γάμοι μεταξύ, διαφορετικών μεταξύ των υπηκών διαφορετικών κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το 2012 θα παρουσιάσει μια έκθεση και σχετικά στατιστικά στοιχεία για την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη του κανονισμού 2001-2002, τον λεγόμενο Βρυξέλλες 2. Ε, η έκθεση θα περιλάβει και τον αριθμό των απαγωγών ανηλίκων, ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε διαρκή άνοδο. Μεταξύ άλλων, επανερχόμενοι στον ρόλο της διαμεσολάβησης, ε, θα ήθελα να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη το 1987 είχε εντοπίσει ε, στον θεσμό της διαμεσολάβησης μια πιθανή εναλλακτική ε, λύση επίτευξης κάποιας συμφωνίας μεταξύ γονέων, μεταξύ ενηλίκων, ιδίως όταν ε, ε, υπάρχει ένας ανήλικος. Στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το πρόγραμμα του 2009, υπάρχουν κάποιες πολύ σαφείς ενδείξεις ακριβώς για τα θέματα αυτά. Στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης ε, γίνεται αναφορά για μια αυξημένη, εντυνόμενη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό και γίνεται και αναφορά στην οικογενειακή διαμεσολάβηση σε διεθνές επίπεδο. Το ίδιο το Συμβούλιο αναφέρει ότι όσο αφορά την απαγωγή ανηλίκων απογονείς, πέρα από την εφαρμογή των απαραίτητων και εφιστάμενων νομικών εργαλείων, θα πρέπει να διερευνηθεί και η δυνατότητα ε, χρήσης της οικογενειακής διαμεσολάβησης σε διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τις ορθές πρακτικές, βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν στα κράτη-μέλη. Το ζήτημα της διαμεσολάβησης λοιπόν είναι ένα χρήσιμο, ένας χρήσιμος θεσμός, ο οποίος βέβαια χρήζει περαιτέρω διευκρίνησης και κωδικοποίησης. Τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί αυτό το αξίωμα του διαμεσολαβητή για να ακούσει όλους εκείνους τους πολίτες που εκούσια αναζητούν μια συμφωνία. Ε, ε, μας υποβάλλονται προτάσεις εκ μέρους δύο γονέων συνήθως οι οποίοι λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε το συμφέρον του ποδιού τους θέλουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Σαφέστατα εκεί που είναι δυνατόν βέβαια να επιτευχθεί συμφωνία ε, η διαμεσολάβηση όταν επιτυχαίνει, όταν επιτυγχάνει σίγουρα ανακουφίζει το, ψυχολογικό βάρος ε, και την ταλαιπωρία αλλά και απαλλάσσει τους γονείς από την βαρύγδουπη γραφειοκρατία που συνήθως επιβαρύνει αυτές τις περιπτώσεις αυτό που κάνουμε ως ευρω... διαμεσολαβητές, οικογενειακοί διαμεσολαβητές, δεν είναι να έχουμε μόνο μια καινοτόμα προσέγγιση, η οποία στην... γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ένας πραγματικός ορισμός της διαμεσολάβησης όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, υπάρχουσα νομοθεσία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό που κάνει όταν απευθύνονται σε αυτό δύο γονείς ε, είναι να τους παρέχει μια σειρά από πληροφορίες, να τους παρέχει ψυχολογική στήριξη, να θέσει στη διάθεσή τους το προσωπικό του και του ειδικού του. Ωστόσο στην πραγματικότητα έχουμε περιορισμούς, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός του τι νοούμε, του τι νοείται με τον όρο διαμεσολάβηση. Και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων μας συνήθως δίνουμε, ε, ενημερώνουμε τους γονείς από την αρχή ότι η συμφωνία τους είναι εθελοντική αλλά μπορεί στη συνέχεια να εκτελεστεί με προσφυγή στις εθνικές αρχές τους σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος προφανώς ε, πάντοτε και εξ αρχής ε, ε, εξηγούμε το ρόλο μας, τις αρμοδιότητές μας, αλλά και τα όρια των αρμοδιοτήτων μας. Και, αυτό το εξηγούν οι ειδικοί που συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση. Έχουμε επεξεργαστεί ένα είδος ε, κώδικα δεοντολογίας ε, του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή σε περίπτωση απαγωγής ε, ανηλίκων σε διασυνοριακές υποθέσεις και έχουμε και την οδηγία 2008-52 υπαριθμών 52 που είναι το μόνο κείμενο αναφοράς από νομοθετική άποψη που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, και θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι επί τη βάση του προγράμματος της Στοκχόλμης θα ήταν πολύ ε, χρήσιμο να ενισχυθεί αυτός ο θεσμός της διαμεσολάβησης. Και το ερώτημα που θέτω και στους αρμόδιους ε, επιτρόπους είναι το εξής. Δεν θα ήταν χρήσιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί σε έναν ορισμό ε, να, να, να διευκρινίσει, να εξειδικεύσει ένα νομοθετικό εργαλείο διεθνούς διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές. Να υπάρξει λοιπόν ένας ε, ορισμός ad hoc ε, ενός τέτοιου συστήματος. Ακριβώς για να μπορούμε να έχουμε μια, μια συγκεκριμένη πλαισίωση στο πλαίσιο, σε ένα κανονιστικό πλαίσιο Πού να άπτεται αυτού του τόσο λεπτού ζητήματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρω ότι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, στις αρχές δηλαδή του επόμενου έτους, και η Επίτροπος Ρέντιξ συγκεκριμένα θα υποβάλει μια σειρά από προτάσεις θα παρουσιάσει μια σειρά από προτάσεις για μια πιο ευαίσθητη δικαιοσύνη, πιο ευαίσθητη απέναντι στα παιδιά. Και Πιθανότατα μεταξύ των ε, μέτρων που θα προταθούν θα βρίσκεται και η υλοποίηση, η ενίσχυση του θεσμού της οικογενειακής διαμεσολάβησης, γιατί και αυτός μπορεί να είναι ένας τρόπος ε, κυρίως να αποφύγουμε το να υφίστανται οι ανήλικοι τις χειρότερες συνέπειες ε, του χωρισμού ή του διαζυγίου των γονιών τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ερχόμαστε στη συζήτηση με τους συναδέλφους των Εθνικών ε, Κοινοβουλίων. Ήδη τέσσερις έχουν γυρίσει το λόγο. Μία από την Ολλανδική Γερουσία, από, το Ελληνικό, την Ελληνική Βουλή και δίνω το λόγο πρώτα ή στην εκπρόσωπο του Ολλανδικής Γερουσίας. Κυρία ε, ε, Πρόεδρε, Είμαι μέλος της ε, Ολλανδικής Γερουσίας, ακούσαμε πάρα πολλά και έτσι δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω διότι υπάρχουν ορισμένα θέματα από των οποίων θα ήθελα να κάνω παρατηρήσεις. Μιλήσαμε για τη συμφωνία της Χάγης για την προστασία των παιδιών και ε, υπάρχει ένας ε, δικαστής ε, σύνδεσμος ο οποίος έχει επαφή με τους εθνικούς δικαστές υπάρχει μάλιστα και ένα ειδικό δικαστήριο κατά τρόπον ώστε να υπάρχει και κάποια εμπειρία επί του θέματος και αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ υπάρχει όμως και κάτι το οποίο με ανησυχεί πολύ διότι ε, άκουσα για τις ε, ε, βιολογικές μητέρες και προτού λυθεί αυτό το θέμα θα ήθελα να κάνω μία έκκληση. Θα ήθελα να εξετάσουμε λίγο και την ηθική πτυχή του θέματος αυτού διότι στην Ολλανδία κάνουμε μία, έναν διαχωρισμό. Υπάρχει βιολογική μητέρα κατόπιν υψηλής τεχνολογίας όπου το παιδί δηλαδή έχει ε, έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τα, τις επιθυμίες των γονιών in vitro και μετά έχει εμφυτευθεί στη βιολογική μητέρα που είναι τελείως διαφορετικό από όταν η ίδια η βιολογική μητέρα προσφέρει το γεννητικό υλικό. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις και αν αυτές δεν επιληθούν τότε θα είμαστε πολύ κοντά σε μια κατάσταση όπου ε, ε, ε, πρέπει να συζητήσει κανείς πολύ σοβαρά. Απαγορεύεται στην Ολλανδία να υπάρχει εμπορική βιολογική μητέρα για εμπορικούς λόγους αλλά δεν μπορούμε να, ούτε να το διαπιστώσουμε ούτε να το αποφύγουμε. Άρα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει και μία ιδεώδης δυνατότητα αναπαραγωγού μητέρας πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να εξαιτήσουμε και να ρυθμίσουμε προτού ε, προχωρήσουμε στη ρύθμιση των ε, ε, νομικών πτυχών. Είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ γιατί το παιδί πρέπει να ξέρει από πού προέρχεται. Ενώ εάν ισχύσουν μόνο οι επιθυμίες των γονιών που το εύχονται δεν μπορούμε να περιοριστούμε εκεί. Το παιδί πρέπει να ξέρει από πού θα έρθει και πρέπει να, από πού προέρχεται και πρέπει να έχουμε εξετάσει και τις ιατρικές και τις επιστημονικές πτυχές του θέματος. Επανέρχομαι όμως τώρα στις απαγωγές των παιδιών και οι εμπειρίες μας στην Ευρώπη είναι, είναι αρκετά καλές και μέσω της ε, Συμφωνίας Βρυξέλλες 2 και ε, με τις διεθνείς συνθήκες αλλά έχουμε προβλήματα ε, με την Αμερική γιατί εκεί δεν υπάρχει χρηματοδότηση για τις αγωγές των γονέων ε, υπάρχει όμως ένα πρόβλημα να ρωτιέμαι δεν θα μπορούσε ε, διμερώς η Ευρώπη να συζητήσει με τις Ηνωμένε Πολιτείε για την ε, εφαρμογή του θέματος αυτού. Ευχαριστώ. Θα σημειώσω την πρότασή σας. Η επόμενη η κυρία είναι η κυρία Βασιλική Νόνογλου από την Ελλάδα. Ε, αγαπητή κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνεδροί μέλη της ε, παρούσας ε, συνέλευσης, χαιρετίζω τη σημερινή αξιόλογη πρωτοβουλία και έχω να τονίσω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι, τουλάχιστον σε εμά και όσους είμαστε νομικοί, ότι συχνά εισπράττουμε τη δυσαρέσκεια ότι χανόμαστε στην περιπλοκότητα και στη μετάφραση. Κάπως έτσι τουλάχιστον μας χαρακτηρίζουν. Ε, σήμερα με όλα αυτά τα οποία άκουσα και θα ακολουθήσουν στη συνέχεια πιστεύω ότι μας δίνεται μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα της ε, προστασίας γενικά των ανηλίκων και τη διευκόλυνση της ελεύθερης διακίνησης της οικογένειας και των ανηλίκων βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει κυρώσει πρόσφατα με νόμο του 2009 τη Σύμβαση της Χάγης του 1993 και πιστεύουμε ότι τα κρίσιμα αυτά σημεία της σύμβασης είναι η καθιέρωση εγγυήσεων για την εξασφάλιση της διασυνοριακής υιοθεσίας πάντα προς το συμφέρον του παιδιού με ταυτόχρονο σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματά του η δημιουργία και η καθιέρωση ενός συστήματος συνεργασίας μεταξύ των συμβαλωμένων κρατών προκειμένου να εξασφαλίζονται εγγυήσεις ώστε να αποφευχθούν τα φαινόμενα αρπαγής πώληση αλλά και παράνομης διακίνησης παιδιών. η ελλάδα κινούμενη προς αυτούς τους στόχους ε, συνέστησε μια κεντρική αρχή. Ε, πιστεύω ότι ανεξάρτητα της πολυπλοκότητας της διαδικασίας σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει κάποια κεντρική αρχή διακρατικών υιοθεσιών ώστε να επιτελεί το έργο της κοινωνικής πρόνοιας και έρευνας που αφορά προφανώς, που προσβλέπει μάλλον στο συμφέρον του παιδιού και που αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των ανθρώπων που πρόκειται να υιοθετήσουν, των θετών γονέων. Προφανώς είναι πολύπλοκο και προφανώς είναι δύσκολο το να συγκροτηθεί μια ενιαία κυβερνητική διακρατική ε, πολιτική σε αυτήν την τόσο περίπλοκη και τόσο ευαίσθητη ε, υπόθεση της υιοθεσίας ανηλίκων. Αλλά δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι στην χώρα μου, όπως επίσης και σε άλλες χώρες πιστεύω, υιοθετούνται και ενήλικοι. Είναι πιστεύω ένα κομμάτι που δεν θα πρέπει να διαφύγει του ελέγχου και της ρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι και αυτό ένα στοιχείο που συντελεί στη διευκόλυνση της διακίνησης των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία θα πρέπει να γίνουν και να συζητηθούν, ε, ε, και για την επιτυχία του θεσμού αυτού προφανώς συμφωνούμε στις ε, επισημάνσεις ε, τις οποίες έβγαλε η κυρία ραφαέλα πρελιάσκο και συγχαρητήρια για την εργασία της ότι δηλαδή όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν ακριβή αρχεία επισημαίνουμε ότι εδώ θα πρέπει να τηρηθεί η αρχή της προστασίας των δεδομένων ε, που αφορά βεβαίως όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή άλλης διακρίσεως ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύνολο κανόνων καθοδήγησης και λεπτομερών κατευθυντηρίων γραμμών για την καλύτερη και σωστότερη εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας ότι κάθε μέλος κράτος μέλος ξεχωριστά θα πρέπει να οργανώνει τοπικά προγράμματα αναδοχής και υιοθεσίας ότι θα πρέπει να διοργανώνονται σεμινάρια, καμπάνιες και ούτω καθεξής, να χρησιμοποιούνται επιστήμονες με γνώσεις ψυχολογίας ώστε να διευκολύνουν τις σχέσεις γονέων και τέκνων, όπως επίσης και ότι θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην υιοθεσία ατόμων, παιδιών με ειδικέ ανάγκες. Σε όλα αυτά δεν θα πρέπει να λησμονηθεί ότι είναι απαραίτητο δικαίωμα να διασφαλιστεί και η ακρόαση του παιδιού. Και εκεί απευθύνω ερώτημα ε, στην κυρία Περλιάσκο εάν στην εργασία την οποία έγινε και στις υπόλοιπες κυρίες που προηγήθηκαν μου ε, σε ποιο σημείο θα πιστεύουν ότι θα ε, υπάρχει η οριμότητα ώστε να ζητείται η ακρόαση και βεβαίω το κεφάλαιο που προηγήθηκε για το, δικαίωμα, την θεμελίωση του δικαιώματο ακράσεω, σε ποιο στάδιο, σε ποιο χρόνο ηλικία θα πρέπει οπωσδήποτε να καθιερωθεί υποχρεωτική ακρόαση του ανηλίκου τέκνου, του, του προσιοθεσίαν και επίσης ότι θα πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη προσοχή ε, και βεβαίως είναι ένα θέμα επεξεργασίας φαντάζομαι και αυτό ότι δηλαδή θα πρέπει να γίνει ειδική ρύθμιση όταν θα πρόκειται ο θωτός γονέας ή το τέκνο αντίστοιχα να προέρχεται από χώρες που έχουν εφαρμόσει την ενισχυτική συνεργασία και ε, άλλες οι οποίες δεν την έχουν αποδεχθεί πέραν των γενικών κατευθυντηρίων γραμμών ε, της ε, συνθήκης της χάγης και του κανονισμού των βρυξελών. ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Μανουέλ Αλτάμπα Λαβάλ από την Ισπανική Γερουσία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις πολύ πλούσιες παρουσιάσεις τους. Πρόκειται για ένα από τους κυριότερους πυλώνες του οικογενειακού δικαίου η αναγνώριση της ε, ευθύνης του γονέα και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες από τις σκέψεις μου. Η κοινή επιμέλεια είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό στην Ισπανία. Στη Γερουσία έχουμε πλέον ένα, μια ομάδα μελέτης για να δούμε ακριβώς ε, ποιες είναι οι καλύτερες ε, ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε στον τομέα της κοινή επιμέλειας. Προσπαθούμε δηλαδή να δούμε σε επίπεδο Ισπανίας ποιες είναι οι καλύτερες διατάξεις που θα μπορούσαμε να έχουμε, δεδομένου ότι στην Ισπανία έχουμε ένα από τα πιο ευνοϊκά συστήματα. Δεν ε, πρόκειται για ένα σύστημα που θα μπορούσε αυτομάτως να ε, εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ένας πατέρας ή μία μητέρα δεν θέλει να δει και να ε, περνάει χρόνο με τα παιδιά του, δεν ε, υπάρχει περίπτωση βέβαια να πιέσουμε κανέναν, αλλά πρέπει να έχει κάθε γονέα τη δυνατότητα να το κάνει αν το επιθυμεί. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα της ευθύνης του γονέα και να υπάρχει συμφωνία μεταξύ του πατέρα και της μητέρας προκειμένου να υπάρχει κοινή επιμέλεια των παιδιών. Προσπαθούμε δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερο να διατηρήσουμε την κατάσταση που υπήρχε πριν ε, ε, διαλυθεί ε, ο γάμος. Προσπαθούμε πάντοτε να υπερασπιστούμε το συμφέρον του ανηλίκου. Αυτό συμβαίνει στις περισσότερες νομοθεσίες και η ισπανική νομοθεσία φυσικά δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο πατέρας έχει, έχει στο μυαλό του το συμφέρον του παιδιού του, η μητέρα επίσης, ε, ε, η εισαγγελία, ε, όλοι έχουν στο μυαλό τους αυτήν την ιδέα της, του συμφέροντος του παιδιού. Ο δικαστής όμως θα κληθεί να αποφασίσει ποιο είναι καλύτερο για το συμφέρον του παιδιού. Και θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη ε, απόφαση του δικαστή. Πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να διατηρηθεί το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαφές και με τους δύο γονείς τους, ακόμη και αν εκείνοι δεν έχουν πλέον επαφές μεταξύ τους ε, γιατί ο δεσμός με τον κάθε γονέα εξακολουθεί να υφίσταται και πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Αναζητούμε λοιπόν ένα σύστημα που θα δώσει τη δυνατότητα στους γονείς να συγκεράσουν το χρόνο που αφιερώνουν στη δουλειά τους και στο παιδί τους και αυτό πρέπει να ισχύει και για τον πατέρα και για τη μητέρα του παιδιού. Και πρέπει αυτό να μπορεί να γίνεται ισότιμα, δηλαδή και οι δύο γονείς να μπορούν να ασκούν το επάγγελμά τους και παράλληλα να ασχολούνται με τα παιδιά τους. Αν βεβαίω δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ τους, ο δικαστής είναι εκείνος που θα αποφασίσει. Ο δικαστής θα βασιστεί στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού και ειδικότερα του δικαιώματο διατήρηση επαφών με του γονεί και με του δύο και με τους δύο γονείς. Σε περίπτωση τώρα διασυνοριακού χωρισμού, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα γιατί υπάρχει η κοινοτική νομοθεσία και υπάρχει και η εσωτερική νομοθεσία των κρατών μελών. Άλλωστε, πολλοί ομιλητές έθεσαν το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της ε, συζήτησης και πρέπει η νομοθεσία να δίνει τη δυνατότητα στο δικαστή να μπορέσει να ε, εκδικάσει την υπόθεση όσο το δυνατόν καλύτερα. Μπορεί για παράδειγμα ο πατέρας να ε, πρέπει να μετακινηθεί για να βρει δουλειά κάπου αλλού και ο πατέρας αυτός να έχει την επιμέλεια του παιδιού. Ε, πρέπει να υπάρχει κάθε φορά η δυνατότητα για το δικαστή να βλέπει ποια είναι η πραγματική πρόθεση των γονιών ε, πριν αποφασίσει ε, ποιος θα έχει την επιμέλεια των παιδιών τώρα. Το δικαίωμα της ε, επίσκεψης είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι δύσκολο γιατί ακόμη και η ορολογία δεν είναι η σωστή στην ισπανική νομοθεσία. Μιλάμε για επίσκεψη κάθε φορά που πάμε να δούμε για παράδειγμα έναν γιατρό, έναν δικηγόρο, έναν οδοντίατρο. Είναι μια επίσκεψη. Όμως δεν πάμε να επισκεφθούμε το παιδί μας. Όχι, περνάμε χρόνο με το παιδί μας. Είναι μια στιγμή που τη μοιραζόμαστε με το παιδί μας. Δεν πρόκειται λοιπόν πραγματικά για δικαίωμα επίσκεψης γιατί πάντοτε το δικαίωμα της επίσκεψης αφορά έναν ξένο, έναν άνθρωπο που δεν μας είναι τόσο οικείο. Έτσι έχουν τα πράγματα στην Ισπανική νομοθεσία. Ο όρος ο ίδιο της επίσκεψης μας δημιουργεί πρόβλημα. Τώρα η κοινή επιμέλεια, θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το θέμα γιατί νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί. Υπάρχουν και οι παππούδε, οι γιαγιάδες Όταν διαλύεται ένας γάμος, για παράδειγμα, πρέπει και οι παππούδε να μπορούν να έρχονται σε επαφή με τα εγγόνια τους. Και μάλιστα σε βαθμό περίπου ίδιο με την κατάσταση που υπήρχε πριν από τη διάλυση του γάμου. Θα μπορούσαμε να βρούμε μία λύση στο πλαίσιο μίας ε, προγαμιαία συμφωνίας, η οποία θα έπρεπε να γίνεται σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Εμείς προσπαθούμε να το επεξεργαστούμε αυτό το θέμα στην Ισπανία, προσπαθούμε να λύσουμε με τέτοιο τρόπο το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ. Και πάλι σχετικά με το δικαίωμα επίσκεψης και επαφής ε, με το, ε, ε, με το παιδί είναι ένα θέμα μετάφρασης και πρέπει να μιλάμε για δικαίωμα επίσκεψης, όχι επαφής όπως είναι ο γερμανικός όρος επικοινωνίας. Ε, βεβαίως ε, αυτό οθεί τους περισσότερους γονείς να συνάψουν μία συμφωνία αλλά ε, ε, ο αριθμός των ατόμων ε, που, ε, έχουν ένα προγαμιαίο συμβόλαιο αυξάνεται τώρα στην Γερμανία και επίσης η επιμέλεια είναι, διεξάγεται από κοινού. Και τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Ντεσέβα από την ε, Επιτροπή, Επιτροπή του Κοινοβουλίου να παρέμβει. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσει θα ήθελα να κάνω στους ε, ομιλητέ Είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε την απάντησή τους, παρά το γεγονός ότι γνωρίζω ότι ο χρόνος μας ε, δεν είναι με το μέρος μας. Στο άρθρο 13 της Σύμβασης της Χάγης αναφέρεται αυτό το ζήτημα της βίας. όσον αφορά την επιστροφή στο χώρο όπου είχε ασκηθεί η βία. Συνήθως οι άντρες την ασκούν, αλλά μερικές φορές την ασκούν και οι γυναίκες. Τα παιδιά λοιπόν είναι στο επίκεντρο αυτές της ίδιας, αυτής της βίας. Και τι γίνεται στην περίπτωση λοιπόν της κοινή επιμέλειας ε, και από την άλλη Ποια είναι η δική σας εμπειρία σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 13 σε περίπτωση ε, οικογενειακής βίας. Το δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω για τους τρεις πρώτους ομιλητές ε, της απογευματινής συνεδρίας. Μιλήσαμε για το άρθρο 46 και για την πρόταση κανονισμού για τα ζητήματα διαδοχής. Μιλήσαμε επίσης ε, για το μιλήσαμε για το άρθρο 46 και σήμερα το απόγευμα οι πρώτοι ομιλητές επανήλθαν στο ζήτημα αυτό και, για τη, στη δικαστική συνεργασία επί του θέματος. βασιζόμαστε στις γνώσεις που έχουμε, γιατί πρέπει να σας πω ότι στα Κανάρια νησιά ετέθη το ζήτημα. Έγιναν σημαντικές προσπάθειες. Ε, μερικές φορές ε, το αποτέλεσμα δεν ήταν το κατάλληλο και ενδεχομένως μερικές φορές να μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτή τη γνώση της κατάστασης που έχουμε για να μην δημιουργήσουμε περαιτέρω προβλήματα. Όταν δύο ενήλικες το επιθυμούν, το διαζύγιο είναι πιθανό. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να αναζητούμε και άλλους λόγους για το διαζύγιο. Δεν υπάρχει λοιπόν ε, ένα δικαίωμα επίσκεψης, υπάρχει ένα χρέος επίσκεψης για να το πω έτσι. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής ε, αν δεν υπάρχει ενοχής και αν, αν δεν υπάρχει ενοχή και αν ε, ε, είναι κοινή συνενέση το διαζύγιο, ε, τότε μπορεί να έχουν κοινή επιμέλεια οι γονεί των παιδιών, εκτό εάν ε, αποδειχθεί ότι αυτό αντίκειται στο συμφέρον του παιδιού, δηλαδή το να βρίσκεται με τη μητέρα του ή με τον πατέρα του. Πρέπει όμω αυτό να αποδειχθεί τη στιγμή τη εκδίκαση τη υπόθεση. Δεν νομίζω λοιπόν ότι έχει νόημα να χρησιμοποιούμε επιχειρήματα που ε, καθιστούν την κατάσταση πολύ πιο περίπλοκη λέγοντας ότι ο ένας γονιός είναι καλύτερος από τον άλλον. Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις επαφές μεταξύ των γονέων και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε ολόκληρη τη δικαστική διαδικασία και την παρέμβαση του δικαστή. Έχουμε μία δικαστική κουλτούρα. Υπάρχουν βέβαια διάφορες συνιστώσεις, η γερμανική συνιστώσα, η πιο λατινική συνιστώσα. Ε, έχουμε όμως και μία κοινή ε, προσέγγιση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να ισχύσει, δηλαδή μια τέτοιου είδου στάση, μια τέτοιου μια τέτοια νοοτροπία σε σχέση με τα δικαστικά, με τα νομικά συστήματα των άλλων κρατών μελών. Αν μόνο εγώ όμως το λέω αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ένα δικαστικό σύστημα, ένα νομικό σύστημα για το οποίο, στο οποίο μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Έχουμε κάνει πάρα πολύ προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο ασφάλειας και δικαιοσύνης. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε διάφορες απόψεις για διαφορετικά μοντέλα και να λέει ο καθένας ότι είναι καλύτερος από τον άλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φραντσέσκα Αλμάιντα από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου για τη συνεδρίαση αυτή ήταν πραγματικά ιδιαίτερος ενημερωτική για μας. Ξέρω ότι υπάρχει πίεση χρόνου, οπότε θα ήθελα να θέσω ορισμένα σημεία σε σχέση με τις ομιλίες που άκουσα. Για παράδειγμα, το θέμα των διασυνοριακών ε, διαφορών. Καταρχάς, η αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων άλλων κρατών μελών σε σχέση με την ε, γονική ευθύνη. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια να ακούσουμε το παιδί και θα έπρεπε να υπάρχει μια υποχρέωση ακρόασης του παιδιού, ειδικότερα όσον αφορά τα ζητήματα ευθύνη του γονέα. Όμω, όπως ακούσαμε σήμερα, υπάρχουν διαφορετικές διατάξεις, διάφοροι τρόποι να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ακρόαση του παιδιού και νομίζω ότι Φοβούμαι ότι μπορεί να οδηγήσει σε μια αδυναμία αναγνώρισης των αποφάσεων ε, ε, σε σχέση με την ευθύνη των γονέων από ένα άλλο κράτος μέλος. Γιατί κάποιο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι δεν έγινε σωστή ακρόαση του παιδιού σε ένα άλλο κράτος μέλος όπου ελήφθη η απόφαση. Οπότε το ερώτημα είναι το εξή. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές για την διαδικασία της ακρόασης ε, των τέκνων, ώστε να μην δημιουργηθεί εμπόδιο στην αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και φυσικά να μην οδηγηθούμε σε τεράστιες καθυστερήσεις στις νομικές διαδικασίες, κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι ούτε για το παιδί. Τώρα για τη διεθνή υιοθεσία. Το συμφέρον του παιδιού είναι το σημαντικότερο στοιχείο ε, στη διαδικασία υιοθεσία στην Πορτογαλία. Γίνεται πάντοτε μια προσπάθεια εξέβρεση τη καλύτερη δυνατή οικογένεια για το παιδί. Το αποτέλεσμα δεν είναι πάντοτε βέβαια αυτό που θα ε, επιθυμούσαμε. Υπάρχει μάλιστα και νέος νόμος ε, σε σχέση με την υιοθεσία παιδιών που έχουν μεγαλώσει σε ένα ίδρυμα, για παράδειγμα. Αν δηλαδή σε εσωτερικό επίπεδο είναι δύσκολο πράγμα η υιοθεσία, ε, φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι σε διεθνέ επίπεδο, όταν μιλούμε για διεθνή υιοθεσία. Και ειδικότερα όταν κάποιο ταξιδεύει, α πούμε, από το ένα κράτο μέλο σε άλλο. Ειδικότερα όταν υπάρχουν διαφορέ στη διάρκεια τη διαδικασία και προσπαθεί κανεί να συγκεράσει διατάξει διαφορετικών νομικών συστημάτων, στο τέλο δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονό ότι 53, 53 ε, ε, παιδιά μόνο έχουν υιοθετηθεί από Πορτογάλους και 11 παιδιά έχουν ε, υιοθετηθεί από ξένους. Και φαντάζομαι ότι η Πορτογαλία δεν αποτελεί εξαίρεση. Γι' αυτό θα ήταν καλύτερο να έχουμε κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές για τη διευκόλυνση της διεθνούς υιοθεσίας. Αν αυτή είναι η καλύτερη λύση για το παιδί βέβαια. για παιδιά, ας πούμε, κάτω των 12, των οποίων τα αδέρφια έχουν ήδη υιοθετηθεί. Ε, και οι ε, δύο Πορτογάλοι εκπρόσωποι αναφέρθηκαν εις ε, τα θέματα της ακροάσεως του παιδιού και ίσως η εμπειρογνώμων θα μπορούσε να σχολιάσει αν πρέπει να υπάρχει ακρόαση του παιδιού ή όχι. Ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα να αναφέρω κάποια συγκεκριμένη ηλικία. Νομίζω η ηλικία των 7 ή των 8 ετών είναι πολύ μικρή. Στην Σουηδία δεν στέλνουμε καθόλου τα παιδιά στο δικαστήριο αν δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο, 17ο έτος της ηλικίας τους. Θα έλεγα ότι για να εισακουστεί το παιδί στο δικαστήριο, αυτή για μένα δεν είναι η καλύτερη λύση. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να εισακουστεί το παιδί με σωστό τρόπο. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα θέματα θα πρέπει να επιληθούν με άμεση συζήτηση, ιδίω όσον αφορά την υιοθεσία. Ίσως η κυρία Βερδιάσκο μπορεί ε, να τα επιλύσει με τους ενδιαφερόμενους και τώρα δίνω την, ε, στην εκπρόσωπο της Βελγικής Προεδρίας το λόγο για να συνοψίσει. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω ότι είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον απόγευμα. Μιλήσαμε για την γονική μέρημνα, για την προστασία των παιδιών και νομίζω ότι αναφερθήκαμε και σε εθνικές και σε διεθνείς και πάντοτε υπάρχει ευθυξία και ε, συγκινησιακός παράγων. Οπότε ο καθένας αισθάνεται πιο ασφαλής στο, στη δικιά του νομοθεσία όταν υπάρχει μία διένεξη περί των παιδιών μεταξύ των γονιών. Είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς ε, μία λύση που να προστατεύει και τους γονείς και τα παιδιά. Και λόγω της διεθνούς μορφής των σχέσεων γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Άκουσα διάφορα εδώ τα οποία ίσως θα έπρεπε ε, να ε, σημειώσω και να συζητήσουμε και εμείς στη διεύθυνσή μας ε, διότι τα διάφορα διεθνή μέσα που υπάρχουν δηλαδή η συνθήκη Βρυξέλλες 2, 2α έχουν βελτιώσει τις σχέσεις διότι υπάρχει κάποια, κάποιος κάποια ενιαία μορφή και κάποια αυστηρότης. Προχωρά κανείς πιο γρήγορα, επιλύει το θέμα της επιμέλειας και της δυνατότητας επικοινωνίας και ε, υπάρχει, ε, ε, υπάρχει μόνο η δυνατότητα εάν η κατάσταση είναι πολύ άσχημη ε, για ένα παιδί να, παρέμβει, ε, να παρέμβουν οι αρχές. Άρα το θέμα του παιδιού είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη και μετά μιλήσαμε για την, ε, το δικαίωμα κροάσεως του παιδιού, την προστασία του παιδιού, αν το παιδί πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία, σε ποια ηλικία και ηλικία έχει σημασία, άλλοι λένε 7, άλλοι λένε 12 ετών θα το συζητήσουμε και στο Βέλγιο και ίσως αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να σκεφτούμε πώς θα, γίνεται η θα διεξάγεται η ακρόαση των παιδιών, με ποιο τρόπο και θα πρέπει να υπάρξει μία εξειδίκευση ακόμη και των δικαστών αλλά και μία ε, εξειδίκευση για το πού και πόσο θα γίνεται η ακρόαση των παιδιών. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να υπάρχει είτε ένας ειδικευμένο δικηγόρος ή ένα άτομο που μπορεί να παρακολουθήσει το παιδί, να το συνοδεύσει κατά τρόπον ώστε το παιδί να μπορεί να εκφραστεί ήρεμα χωρίς να χρειάζεται να το τραβάνε οι γονείς από τη μια μεριά ή την άλλη και νομίζω ότι εκεί τα διεθνή κείμενα έχουν μεγάλη σημασία. Και σε αυτή τη διεθνοποίηση υλοποίηση ή στα διεθνή συμφραζόμενα των όσων άκουσα Πιστεύω ότι ίσως θα πρέπει να αναπτύξουμε και κοινέ αξίες στην Ευρώπη όσον αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας, ε, την γονική μέρημνα, την ε, γονική ευθύνη, τις ε, οδηγίες, τις αποδεδειγμένες καλές πρακτικές. Θα πρέπει να υπάρξουν ανταλλαγές για τις επιτυχείς εμπειρίες. Υπάρχει η διαμεσολάβηση, η ε, παρακολούθηση σε διεθνές επίπεδο ε, ε, μπορεί ίσως να λύσει κανείς το θέμα νομικά αλλά και διαφορετικά όταν είναι δύσκολη η διεθνής εφαρμογή των διατάξεων αλλά όλοι πρέπει να προασπίσουν τα παιδιά όταν πρόκειται για τα δικαιώματά τους προστασίας ή επικοινωνίας με τους γονείς. Πρέπει όλα αυτά να λυθούν όπως είπαμε διεθνώς σε ένα καλό νομικό πλαίσιο να δοθούν οι αναγκαίες πληροφορίες να μπορούν οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι να έχουν δικαίωμα ε, ε, να αντικρούσουν, να εφεσιβάλουν ε, να είναι ενημερωμένοι για τον τρόπο με τον οποίο οι διενέξεις αυτές επιλύονται ε, είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω και να το προωθήσουμε. Έτσι ολοκληρώσαμε αυτό το, αυτή τη συνεδρίαση για τα δικαιώματα των παιδιών. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη, τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι ε, λύσαμε τα πιο ουσιαστικά προβλήματα, αλλά τώρα θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο Μπερδιγκουέρ, ο οποίος θα προεδρεύσει το τελευταίο σκέλος αυτής της συνεδρίασης. Φτάσαμε στην τελευταία σύνοδο, στην τέταρτη σύνοδο αυτού του εργαστηρίου. το οποίο είναι αφιερωμένο, η τέταρτη αυτή συνεδρία είναι αφιερωμένη στην οικογενειακή κατάσταση. Στην σημερινή συζήτηση για την οικοδόμηση ενός ε, ε, δίκαιου χώρου για τον πολίτη και την οικογένειά του, η αναγνώριση της ε, οικογενειακής κατάστασης είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Προφανώς μπορεί να θεωρηθεί κάτι το περιθωριακό, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό το βασικό δικαίωμα του Ευρωπαίου πολίτη να κυκλοφορεί, να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπιφέρει το δικαίωμα να αναγνωρίζεται στην προσωπική του ταυτότητα, σε όποιο κράτος μέλος και αν ζει ή εργάζεται. Με άλλα λόγια, για τον πολίτη είναι σημαντικό να μπορεί να αποδεικνύει την οικογενειακή του κατάσταση και να του αναγνωρίζεται η εγγραφή ε, των λεπτομεριών του, όπου και αν αυτός διαμένει. Η ελευθερία κίνησης, η ελευθερία κυκλοφορίας δεν μπορεί να διατρανώνεται μόνο, να επιβεβαιώνεται μόνο. Είναι συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της αναγνώρισης της προσωπικότητας. Η ελευθερία αυτή ε, πρέπει διαρκώς να αναγνωρίζεται. Έτσι λοιπόν και το καθεστώς που ισχύει και διέπει τον κάθε πολίτη ε, εμπεριέχει το δικαίωμα του ε, πολίτη να του αναγνωρίζεται εύκολα το δικαίωμα αυτό όχι μέσα από πολύχρονες και περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες αλλά εύκολα και αβίαστα. Αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης δεν πρέπει να θεωρείται φιλοξενούμενος σε άλλο κράτος μέλος. Πρέπει ο ίδιος στην ακαιρεότητα της προσωπικότητάς του να γίνεται δεκτός ως τέτοιος. Αυτό δεν είναι μια παραχώρηση. Δεν πρέπει να, να ντρέπεται για το ότι είναι διαφορετικός από έναν άλλον όσο αφορά την οικογενειακή του κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αναγνωρίζετε αυτό και να εγγυάται κανείς την συνέχεια της νομικής κατάστασης ενός πολίτη όταν αυτός μετακινείται από τη μια χώρα στην άλλη. Και έπειτα Ορίστε, υπάρχουν ένα σημαντικός αριθμός περιστατικών που ανακύπτουν. Πάνω στους χίλιες περιπτώσεις τον χρόνο. Ε, το 1 τρίτο από αυτές τις 5.000 περιπτώσεις ε, εγγραφή στα ληξιαρχεία συμπεριλαμβάνουν διακρατικές πτυχές. Για την, λόγω της έντονης κινητικότητας των πολιτών διαφαίνεται η δυσκολία για την αναγνώριση των συστατικών στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης, των εγγράφων τα οποία ο καθένας κατέχει στην Ευρώπη. Υπάρχουν 80.000 γραφεία ληξιαρχικά στην Ευρώπη. Φοβούμε ότι πολλές φορές υπάρχουν και 80.000 εμπόδια στην εύκολη αναγνώριση, γιατί το κάθε γραφείο έχει τη δική του γραφειοκρατική ε, υπόσταση ε, το πιο εύκολο για, έναν, ε, για το μέλος μιας ληξιαρχικής υπηρεσίας είναι να πει αδύνατον. Ε, αυτό όμως δεν πρέπει να ισχύει στην Ευρώπη, γιατί η ελευθερία της κυκλοφορίας δεν πρέπει να είναι μόνο μια διακήρυξη στα χαρτιά, πρέπει να μεταφράζεται στην πραγματικότητα. Ας σκεφτούμε την ομιμοποίηση ή την μετάφραση των στοιχείων εγγράφων της οικογενειακής κατάστασης και ας πούμε ότι κάποιος πολίτης έχει πολιτιστικές ή οικονομικές δυσκολίες, ότι δεν έχει χρόνο να περιμένει την επίσημη μετάφραση, να υποστεί το κόστος. Τι προσπαθώ να σας πω με όλα αυτά. Ε, επειδή με ενδιαφέρει το θέμα, γι' αυτό δέχτηκα κιόλα να προεδρεύσω εδώ. Είναι κάτι σημαντικό στην καθημερινότητά μας. Να μπορούμε να είμαστε τακτοποιημένοι ως Ευρωπαίοι πολίτες είναι ένα θέμα ίσως όχι τεράστιο με φοβερές διαστάσεις, αλλά αφορά την καθημερινότητά μας και μοιάζει να υπάρχει σημαντική ανισότητα, όπως πάντοτε συμβαίνει στην Ευρώπη, είναι ο πλούτος μας αλλά και η αδυναμία μας. Αυτό φαίνεται να υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην εθνική νομοθεσία όσο αφορά τη μεταγραφή του περιεχομένου των εγγράφων της έγκαμης κατάστασης. Αν μπορεί ένα ζευγάρι να παντρευτεί σε ένα αλφα κράτος μέλος, και θέλει να μετακινηθεί και δεν βρίσκει τα έγγραφα ή δεν μπορεί εύκολα να αποδείξει την κατάστασή του, αυτό γίνεται πρόσκομα στην ελεύθερη κυκλοφορία του. Αυτό δημιουργεί μια περιπλοκή. Γιατί η Ευρώπη πρέπει να περιπλέκει τη ζωή των υπηκών τη, Γιατί συνεχίζουν τα κράτη-μέλη να το κάνουν αυτό. Η καταγραφή ενό γεγονότο τη οικογενειακή κατάσταση δημιουργεί μια διαφοροποίηση και μια περιπλοκή. Για παράδειγμα, το επώνυμο. Το επώνυμο. Υπάρχουν χώρες που έχουν ε, θεσμοθετήσει δύο επώνυμα. Άλλες χώρες το αρνούνται και καταγράφουν μόνο το ένα επώνυμο. Α, πολίτες που έχουν διπλή υπηκότητα έχουν στο ένα διαβατήριό τους στο ένα επιθετό τους, στο άλλο διαβατήριό τους στο άλλο επιθετό τους. Όλα αυτά δημιουργούν δυσκολίες ακόμα και στην άσκηση των δικαιωμάτων τους γιατί δεν είναι αναγνωρίσιμοι ως φορείς των δικαιωμάτων τους το δικαίωμα στο όνομα είναι το δικαίωμα στην ίδια μας την υπόσταση. Πρέπει να γίνεται αναγνωρισμένο από όλου το όνομα που εμείς θέλουμε, όχι το όνομα που η νομοθεσία θέλει. Είναι λοιπόν πράγματα που άπτονται της καθημερινής ζωής των πολιτών μας. Και υπάρχουν τεράστιες ανισότητες στην ρύθμιση του γάμου. Δεν υπάρχουν μόνο τα κλασικά ζητήματα της ομοφιλοφιλίας ή ετεροφιλοφιλίας αλλά ε, ε, πάρα πολλές πτυχές του θεσμού του γάμου δεν συμπίπτουν ε, από τη μία χώρια στην άλλη και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα τουλάχιστον για όσο αφορά την διαπίστευση, την πιστοποίηση και την αναγνώριση και υπάρχουν και, συνα... και... δυσκολίες οι οποίες συνδέονται με, τις... τα διαφορετικά συστήματα των κρατών μελών και αυτό τι δημιουργεί εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να ενσκύψουμε στο πρόβλημα και υπενθυμίζοντα τη συμπεριφορά άλλων θεσμών και οργάνων. Ε, οργάνων που ασχολούνται με την επίλυση πρακτικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες λόγω των διαφορετικών διοικητικών και νομικών ρυθμίσεων. Στι 25 Νοεμβρίου του 2009 στην έγκριση του προγράμματος της Στοκχόλμη συζητήθηκε από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ε, τα δικαιώματα τη Ευρωπαϊκή Υπηκότητα. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε και να επιλύσουμε το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης των εθνικών ε, εγγράφων της οικογενειακής κατάστασης. Αυτό ε, αναπαριστά μια σημαντική ιδεολογία. Την αναγνώριση των δικαιωμάτων, την αναγνώριση των τίτλων σπουδών και την αναγνώριση των στοιχείων της οικογενειακής μας κατάστασης. Είναι διαφορετικές πτυχές του ίδιου πράγματος. Δεν είναι ότι θέλουμε μια ενιαία ομοιόμορφη νομοθεσία. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Θέλουμε να υπάρχουν και να πληρούνται οι προϋποθέσεις μιας αμοιβαία εμπιστοσύνης, μιας αμοιβαία αναγνώρισης. Εάν κάτι κάνει ένα κράτος μέλος που δεν αρέσει σε ένα άλλο κράτος μέλος και για το λόγο αυτό παρεμποδίζει την κινητικότητα των πολιτών, αυτό δεν είναι σωστό. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει μια ενδιαφέρουσα πράσινη βίβλο που θα προάγει το δικαίωμα στην μεταγραφή, την ε, αλλαγή και την ταχύτητα με την οποία διεκπεραιώνονται οι σχετικές ε, διαδικασίες που αφορούν τον Ευρωπαίο πολίτη. Εμείς πρόσφατα εγκρίναμε μία έκθεση που παρουσιάστηκε στο Κοινοβούλιο για το πλάνο εφαρμογής του προγράμματος της Στοκχόλμης. Και ένα, μία από τις δράσεις που προτείνονται είναι ο σεβασμός των απαιτήσεων και των επιταγών των πολιτών. Στο 88% οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν απαραίτητη την εφαρμογή μέτρων που προτείνει το ευρωμαρόμετρο, έτσι λέει το ευρωμαρόμετρο, ε, μέτρων ε, αμεβαίας αναγνώρισης των λεπτομεριών της οικογενειακής τους κατάστασης. Είναι ένας ε, στιχ... Ο στόχος λοιπόν είναι μια κοινή απάντηση στο πρόβλημα που να εγγυάται στους πολίτες ένα ισοδύναμο επίπεδο Προστασία των δικαιωμάτων τους όπου και αν βρίσκονται, ιδίω όσο αφορά το δικαίωμά τους στην ταυτότητά τους, στο όνομά τους, στο δικαίωμά τους να τα ασκούν και να τα χρησιμοποιούν, το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή τους και το δικαίωμα στον ε, γάμο τους και στις σχέσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξυπηρετεί τον πολίτη. Αυτός είναι ο στόχος τον οποίο θέλουμε να υπηρετήσουμε ο εθνικός εγωισμός δεν μπορεί να αποτελεί εμπόδιο. Η ανισότητα των εθνικών κανονισμών και νόμων δεν πρέπει να δημιουργούν δυσκολίες στην ελεύθερη διακίνηση των προσώπων και πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη στα νομικά συστήματα των άλλων κρατών μελών. Και αυτό πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση και στην αμοιβαία κατανόηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια, εξού και αυτή η πρωτοβουλία, και τα Εθνικά Κοινοβούλια λοιπόν πρέπει μαζί με την κοινωνία των πολιτών να διεξάγουν έναν κοινό διάλογο πάνω στο θέμα αυτό. Και με αυτές τις σκέψεις ε, θέλω να ανοίξω τη συζήτηση, ε, να παρουσιάσω τους ειδικού μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μας παρουσιάσουν ε, θα μας παρουσιάσει η Επιτροπή της επιδιώξης της για την Πράσινη Βίβλο και θα μας παρουσιάσει τις προσπάθειές της για τη διευκόλυνση της διακυβερνητικής συνεργασίας. Ο χρόνος ε, για όλους τους ομιλητές περιορίζεται σε 10 λεπτά. Τώρα θα δώσω το λόγο στον καθηγητή Πολ Λαγκάρντα, ε, καθηγητή δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Ο τίτλος της παρουσίασής του είναι η αναγνώριση και καταγραφή των εγγράφων οικογενειακής κατάστασης σε διασυνοριακές περιπτώσεις, η υφιστάμενη κατάσταση στα κράτη-μέλη και οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ, καθηγητά Λαγκάρτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως το είπατε και εσείς στην αρχή, το δικαίωμα κάθε πολίτη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαβεί ε, και να διακινείται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωρίζεται στην οικογενειακή του κατάσταση, δηλαδή ε, στις πράξεις οι οποίες αποκανίζουν την οικογενειακή του κατάσταση. Πρέπει το άτομο αυτό να μπορεί να διακινείται με τα τα χαρτιά του χωρίς να χάνει ε, την ε, ηθαγένειά του όταν ε, αλλάζει και περνά από τα σύνορα μιας χώρας. Πράγμα το οποίο δεν είναι προφανές τώρα και προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιλύσει το πρόβλημα. Αλλά η Διεθνής Επιτροπή της Οικογενειακής Καταστάσεως η οποία εδρεύει στο Στρασβούργο προσπαθεί με πολύ περιορισμένους πόρους, πολύ λιγότερους από την Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει την αμοιβαία αναγνώριση της οικογενειακής κατάστασης και των σχεστικών εγγράφων και το συμπέρασμα στο οποίο θα καταλήξω επιβάλλεται ε, να συνεργαστούν ε, οι δύο οργανισμοί κατά τρόπον ώστε η ε, Διεθνής Επιτροπή να επωφεληθεί αλλά και να ωφελήσει όλους τους πολίτες μας. Ε, ορισμένες ε, λοιπόν λεπτομέρειες. Όταν κινείται κανείς και ταξιδεύει μαζί με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα πρέπει να μπορεί να ε, αποδείξει την ταυτότητά του όταν ε, διακινείται και εξασκεί το δικαίωμά του ελεύθερης διακίνησης. Θα πρέπει να αναγράφονται και τα ε, διάφορα, οι διάφορες αλλαγές της οικογενειακής κατάστασης οι οποίες μπορεί να έχουν λάβει χώρα στο εξωτερικό και να αναγνωρίζεται η ηθαγένειά του. Διότι εάν ένα άτομο μεταφερθεί σε μια άλλη χώρα, θέλει να παντρευτεί, να γράψει τα παιδιά του στο σχολείο ή στο τέλος να καταρτήσει το φάκελό του για συνταξιοδότηση, πρέπει να αιτιολογήσει την οικογενειακή του κατάσταση και να βρει ε, έγγραφα τα οποία ενδεχομένως έχουν ε, καταρτιστεί στην ε, χώρα του προέλευσης. Και θα αναφερθώ εδώ στη μετάφραση των πράξεων αυτών, διότι ότι στις σημερινές αρχές δεν μπορεί υποχρεωτικά κάποιος να καταλάβει ε, τα έγγραφα κάποιας χώρας της οποίας δεν μιλάει την ε, γλώσσα και δεν γνωρίζει ίσως καν τα οικονομικά στοιχεία. Υπάρχει λοιπόν μία σειρά συμβάσεων για την ε, έκδοση αποσπασμάτων οικογενειακής κατάστασης για να δίδονται στο εξωτερικό κατά τρόπο τρόπον λοιπόν, ώστε κάποιος να μπορεί να τεκμηριώσει το πιστοποιητικό του γεννήσεως γάμου και ούτω καθεξής. Ε, θα πρέπει αυτά τα αποσπάσματα να, ε, να καταρτίζονται σε πολύγλωσσα έγγραφα που αναγνωρίζονται από τις συμβαλόμενες χώρες και η πλέον ολοκληρωμένη σύμβαση από αυτές είναι η σύμβαση υπαριθμών 16 του 1976 σχετικά με τα πολύγλωσσα αποσπάσματα τα, η οποία έχει ε, κυρωθεί μεταξύ άλλων από 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης η κυρία Ρέντινγκ για να επιλύσει αυτό το πρόβλημα προτείνει να υπάρξει ένα ενιαίο έγγραφο οικογενειακής κατάστασης που θα αποδειχνεί την οικογενειακή κατάσταση ενός ατόμου σε οποιοδήποτε πρόβλημα της καθημερινής ζωής. Είναι κάτι το οποίο και η οργάνωση που εκπροσωπώ έχει εξετάσει, το οποίο όμως παρουσιάζει πολλές δυσκολίες εφαρμογής διότι το έγγραφο αυτό θα πρέπει να καταρτιστεί από ισχύουσες πράξεις οι οποίες πρέπει να αναγνωριστούν και δεν πρέπει να επιβαρυνθεί και υπερβολικά κατά τρόπον ώστε στην καθημερινή ζωή, ζωή να μην ε, υπάρξουν μνήες και στοιχεία που δεν χρειάζεται να αερίζονται έτσι ανα πάσα στιγμή. Και ούτως ή άλλως θα χρειαζόταν μια κεντρική εγγραφή όλων των ε, αλλαγών ε, οικογενειακής κατάστασης όταν ένα άτομο ταξιδεύει και αυτό ήταν η δεύτερη προϋπόθεση που έθεσα, διότι ένα άτομο γεννιέται σε μία χώρα, να γνωρίζεται από τον πατέρα του σε ένα δεύτερο κράτος, παντρεύεται σε ένα τρίτο, χωρί σε τέταρτο και ούτω καθεξής. Κάθε φορά υπάρχει μία πράξη η οποία καταρτίζεται για να καταγράψει το γεγονός. Αλλά όταν προετοιμάζεται ένα νέο γεγονός θα πρέπει το κάθε άτομο και ο ενδιαφερόμενος να μπορέσει να αιτιολογήσει όλη την οικογενειακή του κατάσταση και η οικογενειακή ιστορία. Αυτό θα ήταν εύκολο αν όλα καταγράφονταν στο κράτος προέλευσης. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει τώρα, αλλά υπάρχουν πολλές συμβάσεις της οργανώσεώς μου που προσπαθούν να καταρτήσουν μία διεθνή ανταλλαγή πληροφοριών. Δηλαδή, ο ληξίαρχος, ο οποίος καταρτίζει τη ληξιαρχική πράκτη γέννησης ή θανάτου, θα πρέπει να ε, γνωστοποιήσει στον ομόλογο του μια άλλη χώρα, παραδείγματο χάρη της χώρας γεννήσεω του ενδιαφερομένου και για να αναγνωρίζονται αυτέ οι πράξεις και στα δύο κράτη, δηλαδή και από την ε, ε, αρχή η οποία παραλαμβάνει τα έγγραφα, έχουν προβλεφθεί ορισμένα ορισμένα εγγράφων. Βεβαίως είναι ε, ε, πολύ περίπλοκα τα προβλήματα όσον αφορά τις πληροφορίες τις οποίες θα μεταδώσουμε, ποια θα είναι η αρχή αποδέκτης που μπορεί να αλλάζει από τη μια ε, χώρα στην άλλη, πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες, όλα όμως είναι δυνατά και υπάρχει μια διαδικασία για να ολοκληρωθούν. Αυτή η ενημέρωση των γράφων και καταστατικών δεν θα μπορέσει να υπάρξει παρά μόνο εάν υπάρχει πλήρη αναγνώριση και στον, στο κράτος αποδέκτη. Και αυτό είναι το τελευταίο μου θέμα. Δηλαδή η αναγνώριση των πράξεων που τελούνται στο εξωτερικό. Διότι μπορεί κάποιος να μεταβεί σε μία άλλη, ε, σε μία άλλη χώρα με τα έγγραφα τα οποία πρέπει να αναγνωριστούν σχετικά με την οικογενειακή του κατάσταση και όσον αφορά τις δηλώσεις που περιλαμβάνονται ο, ο γάμος, η αναγνώριση, η ε, συμφωνία συμβίωσης θα πρέπει όλα αυτά να αναγνωρίζονται στη χώρα στην οποία εγκαθίσταται. Και πρέπει να πούμε ότι στο σημείο αυτό άνοιξε δρόμο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αναγνώριση των διαζυγίων. Είναι προφανές ότι ήδη σήμερα μιλήσαμε πολύ για τις Βρυξέλλες 2 ε, Β που επιτρέπουν αυτή την αμοιβαία αναγνώριση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπόρεσε να εκμεταλλευτεί ε, την ιδέα της ευρωπαϊκής ε, ηθαγενείας στην υπόθεση Winking Paul ε, για να καθορίσει το πατρόνιμο ενός παιδιού όπως κατεγράφηκε σε ένα κράτος άλλο από αυτό το οποίο το παιδί γεννήθηκε και διαβεί αλλά πολλά πρέπει που ακόμη να γίνουν διότι τα κράτη γενικώ δεν δέχονται να αναγνωρίσουν μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στο εξωτερικό εάν η κατάσταση αυτή δημιουργήθηκε δηλαδή αναγνωρίζουν την κατάσταση αυτή μόνο εάν έχει τελεστεί σύμφωνα με το ε, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο το οποίο το κράτος θεωρεί ως εφαρμόσιμο. Για να διορθωθεί η αναγνώριση την οποία απαιτούν πολλοί ενδιαφερόμενοι θα έπρεπε να μην υπάρχει πλέον συμμόρφωση στον ε, κανόνα της ε, διαμάχης του Φόρουμ ε, Λόκη. Θα έπρεπε λοιπόν να ληφθεί αυτό υπόψη για την αλλαγή φύλου, για την αλλαγή ονόματος και για τις καταγεγραμμένες συμφωνίες συμβίωσης. Διαπιστώνουμε λοιπόν ένα αποτέλεσμα ατυχές, ότι είναι δύσκολο να διακινηθεί η οικογενειακή κατάσταση, ότι είναι δύσκολο να καταγραφούν τα γεγονότα που τελέστηκαν ή στο εξωτερικό και ε, γι' αυτό θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε ε, τις, ε, την έμπειρη γνώμη της, του αρμοδίου οργανισμού και αυτό μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους. Καταρχήν θα μπορούσε το κράτος να χρησιμοποιήσει το καλύτερο έγγραφο της Διεθνούς Επιτροπής για την Οικογενειακή Κατάσταση ε, και ε, να καταρτήσει ένα νομικό έγγραφο οπότε θα μπορούν να παρακολουθηθούν και υπεραιτέρω περαιτέρω πράξεις μετά θα μπορούσε να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να κυρώσουν ορισμένες συμβάσεις της ICCS και όσον αφορά την, την έκδοση των πολυγλωσσικών πιστοποιητικών θα μπορούσε να ισχύσει αυτό και η τρίτη δυνατότητα θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει ή στις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της CEC, ε, e e, δηλαδή της ICCS, όπου δεν προβλέπεται οικονομική ε, οικονομική ε, ε, ε, ρύθμιση αλλά τίποτα δεν εμποδίζει αυτό να μπορέσει να γίνει. Και εδώ αναφέρομαι στις προσωπικές μου απόψεις χωρίς όμως να αναφερθώ στον οργανισμό στον οποίο συμμετείχα εδώ και πολλά χρόνια. Δεν νομίζω ότι πρέπει να προτιμήσουμε τη μία μέθοδο ή την άλλη αλλά πρέπει να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να τα συνδυάσουμε προς όφελος των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ καθηγητά Λαγκάρτα. Και τώρα ο λόγος ε, στην Σαντάλ Νάστ, Διευθυντή της Διεθνούς Επιτροπής για την Οικογενειακή Κατάσταση. Oui, merci, ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο μετά από τον κύριο Λαγκάρντ. Ε, θα επαναλάβω μερικά από όλα όσα είπε. Αλλά θα ήθελα καταρχάς να πω ότι το να παρουσιάσω σε μερικά λεπτά τις εργασίες ε, της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης ε, στο εξής ΣΥΕΚ είναι σχεδόν αδύνατον. Η καταχώρηση των ονομάτων ε, είναι ένα παράδειγμα, είναι κάτι για το οποίο δούλεψε πάρα πολύ η ΣΥΕΚ και έχει σημασία στο πλαίσιο όλων όσων συζητούμε σήμερα, όμως ε, εκπροσωπεί δυστυχώς τον ξένο στο πλαίσιο αυτών που μου ζητήθηκε να αναλύσω, οπότε θα επικεντρωθώ στα δύο άλλα σημεία. Δεν θα παρουσιάσω επίσης ε, πάρα πολύ την ΣΥΕΚ, γιατί ο κύριος Λαγκάρντ ανέφερε ορισμένα πράγματα για τη Διεθνή Επιτροπή Προσωπικής Κατάστασης κατάστασης, όμως θα ήθελα να σας παραπέμψω στο γραπτό κείμενο το οποίο σας διενεμήθη προηγουμένως και το οποίο είναι πολύ πιο πλήρε σε σχέση με ε, την ΣΥΕΚ, αλλά όπως επίσης και σε σχέση με τα θέματα που θα αναπτύξω. Υπόθηκε ήδη ότι η ΣΥΕΚ έχει δύο κατηγορίες. Εναρμόνιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων και των οικογενειών και αναγνώριση ορισμένων ζητημάτων που είναι πιο τεχνικά, ε, εγγράφων που αφορούν ειδικότερα πιο τεχνικά ζητήματα, ληξερχικές πράξεις ε, ή ε, πρόβλεψη ληξερχικών πράξεων που προορίζονται για το εξωτερικό. Γι' αυτά θα ήθελα να σας μιλήσω σήμερα. Είναι, είναι, δεν είναι σημαντικό για κάποιο κράτος μέλος να είναι ίδιοι νόμοι σε όλα τα κράτη-μέλη, γιατί αυτό που ενδιαφέρει το κάθε πρόσωπο είναι αν μένει στο εξωτερικό και αν του ζητήσουν ε, μία ληξιαρχική πράξη, για παράδειγμα, να μπορεί να λάβει από τις αρμόδιε εθνικές αρχές ένα τέτοιο έγγραφο και να γίνεται αποδεκτό χωρίς ε, πολλές ε, Διαδικασίε στο χώρο διαμονής τους, στη χώρα διαμονή τους. Δηλαδή, αν κυκλοφορούν ε, οι πολίτες, ε, πρέπει και όλα τα έγγραφα που τους αφορούν να μπορούν και αυτά να κυκλοφορούν. Και το είπατε και εσεί στην εισαγωγή σας, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό το δικαίωμα κυκλοφορία δεν πρέπει να είναι απλώς ε, μία δήλωση. Στο πλαίσιο τη ΣΥΕΚ δεν είναι μία απλή δήλωση, γιατί αυτή είναι η αρχή βάση που εφαρμόζει η ΣΥΕΚ εδώ και 60 χρόνια. Οπότε για να διευκολύνουμε την διεθνή κυκλοφορία των ληξιαρχικών πράξεων αλλά και την κατανόησή του στο εξωτερικό, η ΣΥΕΚ e e έχει ε, πρόσβαση σε διάφορες συμβάσεις ε, οι οποίες ε, είναι ή κωδικοποιημένες ή πολύγλωσσες. Σε όλες τις περιπτώσεις, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, τα έγγραφα αυτά δεν χρειάζεται να μεταφραστούν ή να επικυρωθούν ή να περάσουν οποιαδήποτε διαδικασία και γίνονται αποδεκτές ε, ως αποδεκτικό στοιχείο σε άλλες χώρες. Τώρα, ε, αυτό παρουσιάζεται στο παράρτημα 4 ε, σε, ε, σε, πολλές, ε, σε πολλά έντυπα πολύγλωσσα. Δίνουν δηλαδή τη δυνατότητα κάποιων εντύπων που είναι προμεταφρασμένα και έχουν και συγκεκριμένα νούμερα και απευθύνονται στις ξένες αρχές. Όταν γίνουν πάρα πολλές οι γλώσσες, η ΣΥΕΚ, η ίδρυσε e e ένα νέο σύστημα για την, μετα... για την αντικατάσταση του μεταφρασμένου εντύπου με ένα εντύπο με αριθμούς. Στο άρθρο 4 αναφέρονται διάφοροι τρόποι, πώς, πώς μπορούμε δηλαδή από τη, βάση ενός συγκεκριμένου μοντέλου εγγράφου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό σε περιπτώσεις διεθνούς κυκλοφορίας. Το μοντέλο, το πρότυπο εγγράφου είναι το πολύ σημαντικό, ε, ειδικότερα η Σύμβαση 16 της Βιέννης του 1976, το είπε και ο κύριος Λαγκάρτ προηγουμένως, και η οποία ισχύει ε, για 20 κράτη αυτή τη στιγμή. Η Σύμβαση Παριθμών 10 πράξη προβλέπει διεθνή μοντέλα ληξιαρχικών πράξεων γάμου, θανάτου, γέννησης ε, και επίσης μπορούμε να αναφερθούμε και στο πολύγλωσσο μοντέλο των ε, ε, πιστοποιητικών δυνατότητα σύναψης γάμου, τη σύμβαση του 1980 που επιτρέπει να γίνει ένας γάμος στο εξωτερικό. Αυτή η σύμβαση υπάρχει από το 1980 και αυτό το πιστοποιητικό αυτή τη στιγμή ε, παρέχεται ε, σε 10 χώρες. Η αναθεώρηση του, της ορολογίας που χρησιμοποιείται στα παραρτήματα έχει ξεκινήσει για να ληφθούν υπόψη οι εθνικές νομοθεσίες οι οποίες ε, έχουν επιτρέψει τους γάμους ατόμων ιδίου, ιδίου φύλου. Υπάρχουν διάφορες λίστες με παραδείγματα και σας παραπέμπω στη Σύμβαση 17 του 1977 που αφορά την κατάργηση υποχρέωσης επικύρωσης ορισμένων ε, ε, εγγράφων και ισχύει εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι μια ευρύτερη σύμβαση γιατί προβλέπει κατάργηση υποχρέωσης επικύρωσης για όλα τα έγγραφα και τις πράξεις που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση, ε, για την οικογενειακή κατάσταση φυσικών προσώπων, για την ηθαγένειά τους, την εθνικότητά τους, τον τόπο διαμονής τους ε, και παραθέτω το άρθρο το σχετικό και για οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που προβλέπονται για την ε, σύναψη γάμου ή την απόδειξη οικογενειακής κατάστασης. Ε, πρόκειται λοιπόν για έναν τρόπο ελέγχου, ε, παλήθευσης του συγκεκριμένου εγγράφου, της γνησιότητας του εγγράφου, μέσω μιας, ενός εγγράφου, εγγράφου που έχει καταρτιστεί σε πολλές γλώσσες. Υπάρχει και ένα, ένα πρόγραμμα ηλεκτρονική πλατφόρμα, ε, το οποίο είχε ω αποτέλεσμα πολλέ συζητήσει, ειδικότερα για οικονομικού λόγου. Ε, είναι ένα αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο σκοπό έχει να χρησιμοποιήσει τι νέε τεχνολογίε για την κυκλοφορία των ε, ληξιαρχικών πράξεων. Βέβαια αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των εργασιών τη ΙΕΚ και θα διευκολύνει τη ζωή των πολιτών και των οικογενειών και στην Ευρώπη αλλά και εκτό Ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή ε, Δηλαδή θέλουμε μία πλατφόρμα ανταλλαγή ε, μέσω τη ηλεκτρονική οδού ε, των ληξιαρχικών πράσεων. Το 2008 έγινε ένα πρωτότυπο για να δούμε, να δοκιμάσουμε την, ε, το πόσο εφικτό ήταν το πρόγραμμα αυτό. Το πρωτότυπο αυτό ε, άρχισε να ισχύει από το Μάρτιο του 2009 με επιτυχία. Εν τω μεταξύ όμως ε, η ΣΥΕΚ έλαβε συγχρηματοδότηση χρηματοδότηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την αστική δικαιοσύνη και τα διακρατικά προγράμματα. Στην αρχή ήταν ένα εργαλείο επικοινωνίας, ε, ε, ε, υποκαθίσταται η ταχυδρομική θηρίδα από κάποιο άλλου είδους θηρίδα, ηλεκτρονική, και μετά από μία πρώτη περίοδο ανάπτυξης του προγράμματος, όπου περιορίστηκε στην μεταφορά εγγράφων ε, ε, συμβάσεων στα οποία ε, έχει προσχωρήσει ένα, κράτος, ένα κράτος μέλος άρχισε να ισχύει σιγά σιγά και για διμερείς συμφωνίες αλλά και για ανταλλαγές πληροφοριών εθνικών αρχών ακόμη και στην ίδια χώρα και γι' αυτό κάθε κράτος μέλος μπορεί να ε, ε, δημιουργήσει και αυτό τη δική του ηλεκτρονική πλατφόρμα αν δεν το έχει κάνει. Πρέπει να είναι απλό, αποτελεσματικό, ασφαλές ε, και να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα, τα, μικρότερο το κόστος της ιδιότητας του μέλους στην πλατφόρμα αυτή. Μπορείτε να δείτε στο νηστότοπο της ΣΥΕΚ ε, μια ανεπτυγμένη μορφή του συγκεκριμένου πρωτοτύπου. Ο σκοπός είναι να μπορεί να χρησιμοποιείται η πλατφόρμα ανεξαρτήτως του ε, σταδίου που βρίσκεται ε, η μηχανοργάνωση στο, στο κράτος μέλος. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα θέλει απλώς πρόσβαση στο ίντερνετ και τη δυνατότητα του να κινείται κανείς ε, στο ε, ίντερνετ. Για μια απλή και φιλική προς το χρήστη χρήση του συστήματος ε, εμφανίζεται ως ηλεκτρονικό μήνυμα το, το, το έγγραφο που έχει λάβει η συγκεκριμένη αρχή Μόνο όμως ο αποδέκτης, ε, ο παραλήπτης του ε, ε, συγκεκριμένου μηνύματος μπορεί να αποκωδικοποιήσει το συγκεκριμένο έγγραφο και υπάρχει και ένα ελεύθερο κείμενο που σκοπό έχει να δώσει συμπληρωματικές πληροφορίες. Τώρα, τα πολύγλωσσα έντυπα που είναι κωδικοποιημένα και είναι παράρτημα της Επιτροπής ΕΚ που χρησιμοποιούν οι χρήστες συνήθως ε, σε γραπτή μορφή, ε, μεταφέρονται σε PDF ε, και εξαρτάται από τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν ή όχι στη βάση δεδομένων της, την εθνική για να ενημερώσουν τα συγκεκριμένα έγγραφα. Και συμπερασματικά θα ήθελα να σας πω ότι η κατάργηση υποχρέωσης επικύρωσης και μετάφρασης ε, ε, συνιστούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την κυκλοφορία τη διεθνή των πληροφοριών που αφορούν την οικογενειακή, και, την οικογενειακή κατάσταση. Είναι μια σημαντική πρόοδο τόσο για τις εθνικές διοικήσεις αλλά και για τους πολίτες, γιατί σε καθημερινή βάση βελτιώνονται οι σχέσεις τους ε, και με τις αρμόδιες αρχές. Διευκολύνεται η διαδικασία, επιταχύνεται και είναι πολύ μικρότερα και το κόστος αλλά και το χρονικό διάστημα που χρειάζεται αν θα έπρεπε να παρουσιάσουν μόνο εθνικά έγγραφα. Ε, η δυνατότητα λοιπόν ηλεκτρονικής ανταλλαγής τέτοιου είδους εγγράφων θα βελτιώσει την κυκλοφορία των τέτοιου είδους πράξεων ε, και η χρήση των, τεχνολογιών, των νέων τεχνολογιών θα μειώσει πολύ το κόστος. Θα διευκολύνει η πλατφόρμα και θα επιταχύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών και ε, ξένων αρμοδίων αρχών ε, και παράλληλα θα εξασφαλίσει την κυκλοφορία ληξιερχικών πράξεων με πιο ασφαλή τρόπο που δίνει τη δυνατότητα να μειωθεί και να καταπολεμηθεί σε σημαντικό βαθμό ε, η πιθανότητα ε, απατών, παραποίησης ληξιερχικών πράξεων κάτι το οποίο βέβαια είναι ένα φαινόμενο που επιδεινώνεται όλο, όλο και περισσότερο. Ε, ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα αυτό. Ε, η ομάδα μας ε, είναι πραγματικά πάρα πολύ φιλόδοξη, όμως είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία και κατά τη διάρκεια της τεχνικής ανάπτυξης, αλλά και για την, να, το, καταλήξουμε στις ρυθμίσεις που πρέπει να ισχύουν για τη χρήση της. Πρέπει να σας πω ότι οι συμβάσεις ε, στις οποίες ανέφερα είναι ανοιχτά ε, νομικά μέσα και κανένα μέλος ε, δεν αποκλείεται από την προσχώρησή του για να μπορεί να συμμετέχει στη συνέχεια και στην πλατφόρμα αλλαγή πληροφοριών όταν αυτή θα έχει πλήρως αναπτυχθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σαντάλ Νάστ, τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κυρία Σάλα Σάστα Μόινεν από τη Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας σε Πολιτικά Θέματα, Διεύθυνση Α, Πολιτική Δικαιοσύνη, Πολιτικές Διαφορές. Η κυρία Σάλα Σάστα Μοίνεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, από το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα, κρατικά, τα Εθνικά Κοινοβούλια, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη ευχαρίστηση για μένα που βρίσκομαι εδώ και έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω τη μελλοντική πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία δημόσιων εγγράφων και για την αναγνώριση αυτών των εγγράφων. Η πράσινη βίβλος θα υιοθετηθεί στο εγγύς μέλλον το Σεπτέμβριο. Σας μιλώ λοιπόν βάσει των ιδεών που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, αλλά χρήζουν επιβεβαίωσης οι ιδέες αυτές. Είμαι και η τελευταία ομιλήτρια. Ίσως λοιπόν να επαναλάβω ορισμένα πράγματα που ήδη ακούστηκαν ε, στη διάρκεια αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας ημέρας. Ε, την υπομονή σας λοιπόν. Η παρουσίασή μου χωρίζεται σε δύο τμήματα. Καταρχήν θα μιλήσω για τη σημερινή κατάσταση και στη συνέχεια θα παρουσιάσω το περιεχόμενο αυτής της μελλοντικής ε, δημόσιας διαβούλευσης. Καταρχήν γιατί λοιπόν, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα, γιατί ξεκινάει, εγκαινιάζει αυτή τη διαβούλευση για την ε, προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας ε, ε, των δημόσιων εγγράφων και της αναγνώρισης των ληξιαρχικών πράξεων. Νομίζω ότι θα το κατανοήσει κανείς ε, έχοντας συμμετέχει στη σημερινή ημερίδα. Η κινητικότητα των ε, πολιτών είναι μια πραγματικότητα και ενθαρρύνεται από τα δικαιώματα των Ευρωπαίων και προάγεται από τα 20 αυτά εκατομμύρια που μελετούν, εργάζονται και διαμένουν σε άλλα κράτη-μέλη από το κράτος του οποίου είναι υπήκοοι. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι πολίτες στην καθημερινότητα τους αντιμετωπίζουν ακόμη κάποια εμπόδια αναγνώρισης δημόσιων εγγράφων όταν ασκούν τα ευρωπαϊκά τους δικαιώματα. Αυτό τονίστηκε πρόσφατα από την έκθεση της Επιτροπής για το 2010 για την Ευρωπαϊκή Πικότητα. Επίσης επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα του πρόσφατου ευρωμαρόμετρου για τα θέματα πολιτικού δικαίου. Τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων πολιτών είναι υπέρ μέτρων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των δημόσιων εγγράφων μεταξύ των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη και νωρίτερα είχε αναθέσει δύο μελέτες για τον εντοπισμό των προβλημάτων που συναντούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ε, μία για την ε, νομιμοποίηση των δημόσιων εγγράφων και μία για τα αρχικά έγγραφα στα κράτη-μέλη. Και οι δύο μελέτες υπάρχουν στην, ε, στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία από τις πηγές των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι οι απαιτήσει υποβολής στις αρχές των κρατών μελών δημόσιων εγγράφων που να τεκμηριώνουν, να παρέχουν απόδειξη τη έγκαμης, τη οικογενειακής του κατάστασης, έτσι ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν κάποια δικαιώματα ή να αναλάβουν ορισμένε υποχρεώσεις. Τα δημόσια έγγραφα μπορεί να είναι διοικητική φύσεως, συμβολεογραφική φύσεως, ληξιαρχικές πράξεις, συμβάσεις ή δικαστικέ αποφάσεις. Οι πολίτες μπορεί να συναντούν δυσκολίες γιατί τα έγγραφα αυτά δεν γίνονται πάντοτε δεκτά από τις αρχές των κρατών μελών χωρίς τη διεκπαιρέωση κάποιων διοικητικών διαδικασιών όπως η νομιμοποίηση ή η επικύρωση κτλ. Σε αυτή την περίπτωση οι πολίτες ζητούν, κάνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές για την νομιμοποίηση των εγγράφων είναι απαραίτητο να πάει κανείς εκεί αυτοπροσώπως, πόσο θα κοστίσει. Αυτές οι διαδικασίες ε, θα διεκπεραιωθούν σε έμπλοκο χρονικό διάστημα. Χρειάζομαι τα έγγραφα αύριο, θα είναι έτοιμη ε, η μετάφραση αν χρειάζεται μετάφραση. Αυτά μπορεί να φαντάζουν σαν ερωτήσεις ίσονος σημασίας, αλλά δημιουργούν μεγάλη αίσθηση ματέωσης και Δυσφορία στου πολίτε. Μπορεί να μην πάνε στα δικαστήρια οι πολίτε για τα θέματα αυτά, αλλά αυτή η αβεβαιότητα, η ματέωση, ο εκνευρισμό δεν εναρμονίζονται με του ε, στόχους που έχει θέσει η Ευρώπη για τους Ευρωπαίου πολίτε. Όταν μιλούμε για συγκεκριμένα ληξιαρχικά έγγραφα, ένα άλλο ζήτημα ανακύπτει. Και συγκεκριμένα, το ζήτημα της αναγνώρισης των συνεπειών τους, των νομίμων συνεπειών τους, του περιεχομένου τους. Τα έγγραφα αυτά είναι έγγραφα εκδοθέντα από τις επίσημες αρχές του κράτους μέλους που καταγράφουν τα κύρια γεγονότα της οικογενειακής κατάστασης. Γέννηση, γάμος, θάνατος. Όπως ακούσαμε, τα έγγραφα αυτά δεν παράγουν αναγκαστικά τις ίδιες συνέπειες στα άλλα κράτη-μέλη από το κράτος από το οποίο εκδόθηκαν. Κάθε κράτος μέλος έχει τους δικούς του κανόνες για τα θέματα αυτά, τους ίδιους κανόνες ουσιαστικού δικαίου, τους δικούς του κανόνες διεθνούς ιδιωτικού δικαίου, Δικαίου πολιτικής δικονομίας, διαδικαστικούς κανόνες κτλ. Για παράδειγμα, η πατρότητα μπορεί να υπάρχει σε κάποιο κράτος μέλος και να βασίζεται σε κάποιο έγγραφο που δεν αναγνωρίζεται κατά ανάγκη σε άλλο κράτος μέλος λόγω των διαφορών μεταξύ των εφαρμοστέων κανόνων. Για να μπορέσουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες και να κάνουμε, και να κάνουμε πιο αποτελεσματική την εξάσκηση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει αυτήν την ε, διαδικασία διαβούλευση για τη μελλοντική πράσινη βίβλο και καλύπτουμε δύο θέματα. Πρώτον, την ελεύθερη κυκλοφορία των δημόσιων εγγράφων και δεύτερον, την αναγνώριση των νομικών συνεπειών των ληξιαρχικών πράξεων. Τα δύο θέματα καλύπτονται γιατί μακροπρόθεσμα στο μέλλον, όπως ακριβώς αναφέρεται και στο σχέδιο δράσης της Στοχόλμης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να εξετάσει την υποβολή δύο νομοθετικών προτάσεων μετά τη λήξη του προγράμματος της Στοκχόλμης. Πρώτον, για την ελεύθερη κυκλοφορία των εγγράφων ε, μέσω της κατάργησης της νομιμοποίησης και δεύτερον, την αναγνώριση των νομίμων συνεπειών ορισμένων ληξιαρχικών πράξεων the public consultation will cover two issues. Για την κατάργηση της επικύρωσης, με συγχωρείτε, των εγγράφων, όχι της νομιμοποίησης. Ε, τώρα, για την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, δημόσιων εγγράφων. Έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ε, γεγονότα απαραίτητα που πρέπει να υποβάλει ο πολίτης στις αρχές. Συχνά οι αρχές απαιτούν επικύρωση μέσω ακριβώς της διαδικασίας αυτής. Και ο στόχος είναι εύλογος. Ο στόχος είναι να αποδειχθεί ότι το έγγραφο είναι γνήσιο και ορθό. Έτσι καταπολεμάται ή προλαμβάνεται μάλλον η απάτη. Πέραν της, μετά την επικύρωσή του το έγγραφο μπορεί να υποβληθεί σε άλλα κράτη-μέλη. Ωστόσο, οι διατυπώσεις στην πράξη αποτελούν φορτίο για τον πολίτη, απαιτούν χρόνο και χρήμα. Όταν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν υπάρχει αυξανόμενη αμοιβαία εμπιστοσύνη στον κοινό χώρο δικαιοσύνης, μια και βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναρωτιέται μήπω θα έπρεπε να καταργήσουμε τη διαδικασία επικύρωσης για όλα τα δημόσια έγγραφα μεταξύ των κρατών μελών. ask. Ε, αυτό απαιτεί τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών και την ανταλλαγή ε, πληροφοριών. Να μπορεί οι αρχές να έρχονται σε επαφή με τις αρχές έκδοσης των εγγράφων αν έχουν κάποια αμφιβολία. Για να επιλύσουμε το ζήτημα της μετάφρασης ή για να μειώσουμε τις μεταφράσεις, εξετάζουμε το ενδεχόμενο τυποποιημένων εγγράφων και είχαμε σήμερα, ακούσαμε τις εμπειρίες από άλλους διεθνείς οργανισμούς που έχουν συντάξει τέτοιες, ε, τέτοια υποδείγματα. Το δεύτερο θέμα τώρα, η αμοιβαία αναγνώριση των νομιμίων συνεπειών των ληξιαρχικών πράξεων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να μαθαίνουμε πάντοτε αν η νόμιμη κατάσταση που δημιουργείται σε ένα κράτος μέλος θα αναγνωρίζεται ή όχι στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Σήμερα έχουμε μία πτυχή που αναγνωρίζεται, το, το διαζύγιο. Αν ένα διαζύγιο έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του κανονισμού Βρυξέλλες 2α, αν ένα άτομο πήρε διαζύγιο στην Ελλάδα, τότε μπορεί να πάει στην Ισπανία και θα ισχύει το διαζύγιο του και θα μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Αυτή είναι μια πτυχή που καλύπτεται, και που καλύπτεται από την αμοιβαία αναγνώριση. Υπάρχουν άλλες πτυχές της οικογενειακής κατάστασης που επίσης μπορούν να γίνονται αμοιβαία αναγνωρισμένες. Η συγγένεια, η αλλαγή του ονόματος που ήδη αναφέρθηκε σήμερα. Τα νομικά συστήματα των κρατών μελών επηρεάζονται από ιστορικά, θρησκευτικά, γλωσσικά και πολιτισμικά φαινόμενα και αυτό είναι κατανοητό. Υπάρχουν λόγοι για τους διαφορετικούς κανόνες της ονοματοδοσίας, για παράδειγμα. Αλλά ε, καταστάσεις όπου οι πολίτες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το όνομα που αντιστοιχεί στην υπηκότητά τους ε, δεν πρέπει να ισχύει ή μπορεί να έχουν διαφορετικά ονόματα οι πολίτες σε διαφορετικές χώρες και αυτά άπτονται της ταυτότητας του ατόμου. Όπως ακούσαμε, έχει γίνει διεθνώς ε, πολλή δουλειά σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση από την Διεθνή Επιτροπή Προσωπικής Κατάστασης. Υπάρχουν και πολλές διεθνείς συμβάσεις, αλλά δεν τις έχουν υπογράψει όλα τα κράτη-μέλη, επομένως δεν έχουν λυθεί ακόμα τα ζητήματα εξ ολοκλήρου. Φυσικά, βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την εμπειρογνωσία της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης στον τομέα αυτό. Και παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τα πιλωτικά τους προγράμματα και για την ηλεκτρονική διαβίβαση των αρχικών πράξεων και εγγράφων. Η πρόκληση λοιπόν είναι να βρούμε τρόπους επίλυσης των προβλημάτων των πολιτών σε σχέση με την αμοιβαία αναγνώριση των ληξιαρχικών πράξεων και η πράσινη βίβλος θα έρθει να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρισκόμαστε στην αρχή της διαδικασίας. Μας ενδιαφέρουν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και ε, θα θέλαμε να ακούσουμε τις απαντήσεις σας ε, στη φάση της διαβούλευσης που θα εγγενιαστεί τον ε, Απρίλιο. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για την διοργάνωση αυτής της πλούσιας ημερίδας. Μας έδωσε πολύ τροφή για σκέψη. Θα μεταφέρουμε αυτά που ακούστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίω για την ανακοίνωση αυτή της διαδικασίας διαβούλευσης. Έχουμε λίγο χρόνο για συζήτηση. Θα θέλαμε να παρέμβουν και οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είναι ευκταίο αυτό, αλλά όχι υποχρεωτικό βέβαια. Όποιος θέλει να λάβει τον λόγο μπορεί να το κάνει. Ερωτώ λοιπόν, θέλει κάποιος να λάβει τον λόγο. Η συνάδελφος Τάινεν. <laughs> Ναι, σαν ε, Ευρωβουλευτήνα θα ήθελα εδώ να παρέμβω και συγχρόνως είμαι Γερμανίδα συμβολεογράφος και μπορώ να σας πω ότι είναι ε, δύσκολη η αναγνώριση των εγγράφων τα οποία είναι αναγκαία για την ε, σύναψη συμβολέων επί διαφόρων θεμάτων διότι καταρχήν χρειάζεται η πιστοποίηση της οικογενειακής καταστάσεως του ακτόμου και αυτό είναι πολύ δύσκολο εάν η απόδειξη και το πιστοποιητικό χρειάζεται πολύ χρόνο για να υπάρχουν σε αποδεκτή μορφή γιατί η Γερμανία είναι μια δύσκολη χώρα που κοιτάζει τον τύπο πάρα πολύ και πολλές φορές χρειάζεται επί χρόνια να ταλαιπωρείται κανείς ε, γιατί δεν έχει τα αναγκαία έγγραφά του ε, και ε, η πείρα μας για τον Καναδά και την Αμερική με τους οποίους είχαμε ε, πολλές συναλλαγές και συμφωνίες που συνήθισαν με Γερμανούς χρειαζόταν προετών χρόνια για να λάβουμε τα στοιχεία ενώ τώρα υπάρχει μια βελτίωση και την οποία χαιρετίζω. Το Ινστιτούτο αυτό που αναφέρατε δεν τον γνώριζα αλλά θα ασχοληθώ έντονα μαζί του και θα έπρεπε σαν ευρωβουλευτές να προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε ως το δυνατόν περισσότερα άτομα, επιμελητήρια για να συνεργαστούμε και να διαβουλευόμαστε περισσότερο πράγμα το οποίο θα διευκολύνει πάρα πολύ την διεκμεραίωση της καθημερινής ζωής των ε, ε, Ευρωπαίων πολιτών και ιδίως όσον αφορά τις επαγγελματικές αυτές τους ε, συμφωνίες και γι' αυτό ευχαρίστως θα ήθελα να καταλήξουμε κάποτε σε μία συμφωνία όπου χώρες σαν την Αμερική, το Καναδά, το Ισραήλ, η Αυστραλία, Αμερική εννοούσα τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλες οι χώρες αυτές ε, να μπορέσουν να μας διευκολύνουν κατά τη σύναψη των συμφωνιών και συμβολέων. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Αναμένω και άλλες αιτήσει ε, λήψεως του λόγου. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε και εμείς μία επιτροπή ε, η οποία συμβουλευτικά επεμβαίνει και θα ήθελα να ξέρω αν ε, η επιτροπή θέλει να έρθει σε επαφή με αυτό το, αυτή την οργάνωση στη χώρα μας. Θέλει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Η καθηγήτρια Μπορώ να απαντήσω στην βουλευτήνα ότι όντως η οργάνωσή μας, η ΣΕΙΕΣΕ, εργάζεται κάπως περίεργα γιατί όταν ένα κράτος γίνεται μέλος οργανώνει ένα εθνικό τμήμα, δηλαδή ορισμένα άτομα τα οποία είναι τα πλέον αρμόδια στον τομέα που ενδιαφέρει την οργάνωσή μας, την ΣΕΙΕΣΕ, και έχουμε εκπροσώπους των Υπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης που ασχολούνται με το θέμα της οικογενειακής καταστάσεως και εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών. Η, οργάνωση λοιπόν σε και ε, το Εθνικό Τμήμα έρχονται σε επαφή ε, με την ε, Ορλανδική οργάνωση που αναφέρατε και ε, πολλοί από αυτούς ε, υπήρξαν ε, μέλη κάποια στιγμή της, του Ολλανδικού Τμήματος της ΕΕΣΕ. Ευχαριστώ, παρακαλώ. Είναι μεγάλη μου τιμή το ότι συμμετέχω σε αυτήν την ημερίδα όπου πρόεδρος είναι η μεγάλη μορφή της Ιταλικής Δημοκρατίας, ο Και είναι μεγάλη μας τιμή κύριε Πρόεδρε το ότι είμαστε πράγματι και εσείς προεδρεύετε αυτό οφείλω να το πω σε εσά. Ε, όσον αφορά τώρα το θέμα της, ε, της διακίνησης των εγγράφων, υπάρχουν πιστεύω ζητήματα που θα πρέπει να λυθούν με ποια έννοια. Ότι τα δημόσια έγγραφα που θα διακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς θα πρέπει να εκτιμηθεί το πόση μεγάλη αποδεικτική δύναμη θα έχουν στο μέλλον σε απόδειξη γεγονότων που δεν χωρεί αμφισβήτησή τους. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κάποια διαδικασία ή να τεθούν οι προϋποθέσεις ώστε τα δημόσια έγγραφα που πιστοποιημένα και επικυρωμένα θα κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι δυνατά σε απόδειξη του γεγονότος εφόσον βεβαίως αποδειγμένα έχουν συνταχθεί από τον αρμόδιο δημόσιο υπάλληλο και έχουν επικυρωθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ αυτό για την επισήμανση της προετοιμασίας της, των δημοσίων εγγράφων της διακίνησής τους και της αποδεικτικής τους δυνάμεως. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ για την συμβολή σας και για την προσοχή σας. Παρακαλώ, είδα και ένα άλλο χέρι. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα και ενημερωτική συζήτηση. Έχω μία ερώτηση να κάνω για τα ληξιαρχικά έγγραφα. Αυτά ισχύουν και για τις ληξιαρχικές πράξεις γάμου. Και τι συνέβη όταν ένα ζευγάρι του ίδιου φίλου παντρεύεται και αναζητεί λεξιαρχική πράξη γάμου και τι αποδεικτική αξία έχει λεξιαρχική πράξη γάμου σε μια χώρα που δεν αναγνωρίζει το γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φίλου και σε σχέση ε, με την πράξη 8133 της συνθήκης Ευχαριστώ για την ερώτηση. Εδώ στα δεξιά μου σίγουρα θα υπάρχει κάποιος που είναι σε θέση να απαντήσει. Πρέγω, πρέγω, Παρακαλώ, κυρία Νάτσα. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά τη μετάφραση αλλά κατάλαβα το τελευταίο μέρος, δηλαδή αν υπάρχουν έγγραφα τα οποία λάμβαναν υπόψη ε, το, τη διαφορετική ορολογία σε περίπτωση γάμου δύο ατόμων του ιδίου φύλου. Ε, στην ομιλία μου ε, τα ανέφερα πολύ γρήγορα αλλά λόγω περιορισμένου χρόνου μίλησα πολύ γρήγορα. Ε, προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να ενημερώσουμε τα έγγραφα τα οποία χρησιμοποιούνται εδώ και 30 χρόνια για να λάβουμε υπόψη την αλλαγή του λεξιλογίου ε, για ε, την σύναψη σχέσεων μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου ή ζευγαριών του ιδίου φύλου, πράγμα το οποίο δεν είναι προφανές έχουμε πρόβλημα ορολογίας, δεν υπάρχει ουδέτερος όρος σε όλες τις γλώσσες γιατί σε ορισμένες χώρες μιλάει κανείς για τον σύζυγο και ε, την σύζυγο ή κάτι τέτοιο στη γλώσσα τους και υπάρχουν και χώρες που δεν γνωρίζουν αυτές τις συνήθειες δεν θέλουν να τις λάβουν υπόψη τους ακόμη και ε, για να αναφερθούν στο λεξιλόγιο για τα έγγραφα. Είναι κάτι το οποίο έχουμε παρακολουθήσει εδώ και πολύ καιρό και φαίνεται ότι ακόμη και τα κράτη τα οποία ήταν τα πλέον διστακτικά για να χρησιμοποιήσουν μία άλλη διατύπωση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε άτομα ανεξαρτήτως φύλου τώρα είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν ε, τα πιστοποιητικά ε, τα πολύγλωσσα ε, βάζοντας νερό στο κρασί τους για τους γάμους και για άλλες σχέσεις. Δηλαδή χώρες οι οποίες ήταν πολύ πλωσιρωμένες στα έγγραφά τους όσο είχαν όπου υπήρχαν παλιές, παλιές διατυπώσεις σύζυγος ή πατέρας, μητέρα διότι δεν ήξεραν ότι μετά από 40 χρόνια θα, υπήρξε, θα υπήρχε νομοθεσία καταργώντας ε, τη χρήση φύλου στο γάμο αρχίζει να βρίσκεται μια λύση όπου πρέπει ε, να ε, υπάρχει ε, μια ένδειξη φύλου καθότι πρέπει να αναφέρεται το φύλο αλλά εάν δεχθούν το, τα κράτη έχουμε βρει μια λύση θα πρέπει όμως να υπάρξει και μια νέα συνθήκη και στη συνέχεια θα πρέπει να κυρωθούν οι συνθήκες αυτές από τα Εθνικά Κοινοβούλιο. Βρήκαμε δηλαδή κατά κάποιον τρόπο μία λύση που μας επιτρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα αλλά στη συνέχεια θα πρέπει να κυρωθεί και βεβαίως σαν εκπρόσωπος της ΕΣΕ πρέπει να σας πω ότι έχω ένα μειονέκτημα σε σχέση με την διπλανή μου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει να περιμένουμε ε, την ε, κύρωση των κρατών μελών και υποθέτω ότι ορισμένοι θα ε, θέσουν προβλήματα σχετικά με όλα αυτά τα οποία είπαμε πολλές φορές για το όνομα παραδείγματος χάρη το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη. Υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν ήταν όσο προοδευτική θα θέλαμε από πλευράς Γενικής Γραμματείας διότι αντιμετωπίσαμε τους δισταγμούς ορισμένων κρατών εν η συνθήκη για την αναγνώριση των ονομάτων ε, δεν είναι τόσο τόσο επίκαιρη διότι υπάρχουν άλλες αποφάσεις αλλά όπως είπε ο κύριος Λαγκάρντ και το διευκρίνησε υπάρχει το θέμα της αναγνώρισης των ε, σχέσεων που ήταν δύσκολο να ολοκληρωθεί αλλά μέχρι στιγμής μόνο ένα κράτο έχει, κράτος έχει υπογράψει, η Ισπανία και η δεύτερη χώρα που την κύρωσε είναι η Πορτογαλία όχι η Πορτογαλία υπέγραψε και ε, η Ισπανία έχει κυρώσει. Άρα δεν έχουμε κάποια λύση η οποία θα επιβληθεί αυτομάτως στα κράτη. Θα ήθελα να προσθέσω από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως εάν η ερώτηση απευθυνόταν και σε εμά για το εάν τα πιστοποιητικά γάμου είναι δημόσια έγγραφα θα ήθελα να πω ότι και τα πιστοποιητικά γεννήσεως και γάμου και διαζυγίου είναι δημόσια έγγραφα και υπάρχουν ουσιαστικοί κανόνες ε, για το, για το γάμο που αναφέρονται ε, στο ουσιαστικό δίκαιο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εφαρμοστούν σε άλλες ε, ενώσεις ή συμβιώσεις ε, αλλά υπάρχει, υπάρχουν οι οδηγίες της ελεύθερης διακίνησης όπου λέγεται ότι ε, το το πιστοποιητικό γραμμού πρέπει να αναγνωρίζει την ελεύθερη διακίνηση ε, για το άτομο που είναι όπως είπα ελεύθερη. Οπότε από δικής μας πλευράς η κατάσταση είναι αυτή και για το μέλλον θα δούμε πώς θα έχουν τα έγγραφα και θα χρειαστεί να δούμε στη συνέχεια ε, εάν μπορούμε να αναλάβουμε αργότερα πρωτοβουλίες. Αλλά η διαβούλευση είναι πολύ ευρεία και μπορούμε να εξετάσουμε διάφορα θέματα. Άλλες, παρεμβάσεις. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή τη συνάντηση. Η συζήτηση έδειξε ότι ήταν ε, σωστή η κίνηση να διοργανωθεί αυτή η συζήτηση και οι προηγούμενες συνεδρίες αλλά και αυτή. Είναι ένα θέμα ιδιάζων, αλλά και σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και συγκεκριμένα το γεγονός ότι τα προβλήματα μιας κοινή απλοποιημένης διαδικασίας ε, των εξιαρχικών πράξεων αποτελούν κομμάτι της ε, ε, κατασκευής της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη και δεν μπορούμε να τα αμελούμε τα ζητήματα αυτά. Οι ομιλητές μας παρουσίασαν όλες τις παραμέτρους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προφανώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διαδικασία που βρίσκεται εν εξελίξη. Αυτή είναι την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης για την πράσινη βίβλο. Τα θέματα που πρότεινε, επικύρωση εγγράφων, να την ε, διατηρήσουμε, να την καταργήσουμε. Ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσει και πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του ζητήματος και καλό θα ήταν να είναι και νομοθετική αυτή η πρωτοβουλία. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης φάνηκε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε έντονες υπερβάσεις, ε, υπό την έννοια ότι θα δώσουμε μία, μία και μόνη ευρωπαϊκή λύση. Η ετερογένεια των εθνικών καταστάσεων, όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, σε όλες τις άλλες καταστάσεις, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να διαφυλαχθεί. Γιατί, Γιατί υπάρχουν παραδόσεις, αλλά και γιατί το θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αρμοδιότητα την οποία δεν μπορεί να υπερκεράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πρέπει να γίνονται σεβαστές οι κοινωνίες. Ωστόσο, το ζήτημα απαιτεί μια κοινή προσπάθεια και η εμπειρία της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης ενισχύει αυτό, αυτήν την προσπάθεια γιατί είναι, μια, είναι κάτι που γεννήθηκε αυθόρμητα από κάτω δεν ήταν μια θεσμική πρωτοβουλία. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεπίδησε από μια ομάδα κρατών και κατάφερε να υπερβεί τις αντιθέσεις. Και μάλιστα ανέκυψε η σχετική ανάγκη και μεταξύ μη ευρωπαϊκών χωρών. Νομίζω ότι και μη ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν σε αυτή τη Διεθνή Επιτροπή. Βεβαίω η αναγνώριση της ληξιαρχική κατάστασης παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα και συνενώνει πολλές φωνές, πράγμα που αποτελεί ενθαρρυντικό δείγμα. Νομίζω επίσης ότι είναι θεμελιώδες να χρησιμοποιήσουμε την μοντέρνα τεχνολογία. Ε, όλοι θυμόμαστε πώς ήταν τα επίσημα έγγραφα οι θηρεοί, οι σφραγίδες ε, που υπήρχαν πάνω σε αυτά τα έγγραφα. Θυμόμαστε ε, τις πρώτες μορφές εκείνων των ληξιαρχικών πράξεων. Έχουμε εμείς οι στο μυαλό μας έτσι τη μορφή του ληξίαρχου. Ε, Ήταν σαν σαν υπήρχε μια ενορία εκεί που ήλεγχε όλα αυτά τα έγγραφα. Αλλά τελικά ε, μέσα από την ενιαία αγορά ξεπίδησε αυτή η ανάγκη ελευθερίας της κυκλοφορίας και της διακίνησης. Είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να δώσουμε τη μέγιστη προσοχή στις προϋποθέσεις και τις συνθήκες αυτές και να εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή το έργο που έχει επιτελέσει η Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Κατάστασης, Οικογενειακής Κατάστασης. Και καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να διευρύνει το περίφημο πρόγραμμα της Στοχόλμης, που αποτελεί ουσιαστικό μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελπίζω ότι και αυτή και αυτή, αυτό το θέμα της πιστοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων θα λάβει την προσοχή που του αξίζει. Εγώ γεννήθηκα στη Σαρδινία θα σας δώσω έναν προσωπικό τόνο. Είναι μια, μια εποχή της Ιταλίας που επί καιρό, όπου επί πολύ καιρό κυριαρχούσαν οι Ισπανοί. Τώρα αποτελεί Ιταλικό έδαφος. Υπάρχουν άτομα που έχουν το, όνομα των οποίων ε, έχουν ισπανική προέλευση και ανέφερε ένα πολύ μακροσκελές όνομα τώρα ο κύριος Μπερλίνγκουερ ε, ένα ένα όνομα που πιάνει σχεδόν μια σελίδα, μπορώ να φανταστώ ότι στο Βέλγιο θα, ήταν, θα δημιουργούσε προβλήματα αναγνώρισης ένα τέτοιο μακροσκελές όνομα. Τι να γίνει, η Ευρώμη απαρτίζεται και από αυτές τις διαφορές. Ποιο είναι το ουσιώδες. Το ουσιώδες είναι ότι πρέπει και να τα σεβαστούμε αυτά, αλλά και να διευκολύνουμε την αναγνώριση και την κυκλοφορία των προσώπων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.